Uh, um, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο, ο κύριος Βαντερ ο πρωταγωνιστής μας, οπότε ε, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Ρούλε και την κυρία Σνάλοβα. Ίσως θα έρθουν και άλλα μέλη εν τω μεταξύ να σας καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας του μηνός Νοεμβρίου. Έχουμε τρεις συνεδριάσεις σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Να ανακοινώσω μία μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. για τη διαθεσιμότητα ε, των ε, ε, ιστοσελίδων των, του δημοσίου θα, θα συζητηθεί νωρίτερα στις 10 και 40 ανάμεσα στις 10 και 40 και 11 και 10 Η ψηφοφορία για την έκθεση Σμιτ θα αναβληθεί για τη 17η Δεκεμβρίου, γιατί η υπεύθυνη επί της ουσίας επιτροπή θα καθυστερήσει και αυτή για θέματα παραβίασης ε, του δικαίου περί ανταγωνισμού και για την εναρμόνιση των μηχανημάτων ε, που λειτουργούν με πίεση θα υπάρξει επίσης καθυστέρηση σχετικά με τη φύση της πρότασης. Θα πρέπει να δούμε αν είναι νέα πρόταση, αν είναι αναδιατύπωση παλαιάς πρότασης. Και έτσι αύριο θα έχουμε ε, περισσότερο χρόνο για τη δεύτερη έκθεση της κυρίας Σενάλοβα. Λοιπόν, με αυτές τις αλλαγές γίνεται δεκτή η διάταξη. Ξέρετε ότι ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Χαιρετώ τους φίλους που μας βλέπουν. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα καινούριο newsletter που κυκλοφορεί επίσης της Επιτροπής μας, το οποίο και αυτό δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει να το παίρνει αυτό με email μπορεί να μας στείλει ένα email στο website του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας πω επίσης ότι είμαστε πιλωτική επιτροπή για συνεδριάσεις χωρίς χαρτιά. Θα παίρνετε δηλαδή όλες, ε, όλα τα έγγραφά σας σε iPad και όποιος ε, θα ήθελε να τα έχει από εδώ και πέρα σε χαρτί θα πρέπει να μας το πει. Προσπαθούμε να είμαστε φίλοι προς το περιβάλλον. Εγκρίνοντας τα πρακτικά της 17ης Οκτωβρίου θα θεωρηθούν δεκτά εκτός και αν τεθεί κάποιο θέμα πριν από το τέλος της συνεδρίασης. Δύο επιπλέον θέματα. Πρώτον, Έχουμε ένα μικρό θέμα για, τον, για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου. Θα μας τις παρουσιάσει η κυρία Σαλντεμόζε, εξ ονόματος της Ιδίας φυσικά και της κυρίας Πιετικάινεν για να μας πει ακριβώς πού βρισκόμαστε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμπορ. Δεν έχουμε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις ε, ακόμη. Περιμένουμε ακόμη το Συμβούλιο. Συζητούν ακόμη κατά πόσο θα δώσουν εντολή διαπραγματευτική ή όχι. Έχουμε βέβαια όλο το πακέτο και το κομμάτι που αφορά την ε, επιτήρηση της αγοράς, αλλά και το κομμάτι που αφορά ε, την ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές. Το πρόβλημα είναι το made in, ε, το που είναι κατασκευασμένο το προϊόν, του διάταξη του άρθρου 7. Έχουμε θέσει κάποιες ημερομηνίες για διαπραγματεύσεις, οποίες αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Ίσως όχι σήμερα, αλλά σε μια-δυο εβδομάδες ε, ελπίζουμε να φτάσει η έκθεση στην Ολομέλεια, γιατί πρέπει να έχουμε ένα, πρόγραμμα και να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε αυτό το σημείο. Ελπίζω ότι κάτι θα καταφέρουμε. Για την ώρα όμως δεν γίνονται διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον όχι μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εντό Συμβουλίου ίσως. Είχα πολλές ε, συνεδριάσεις, συναντήσεις ε, με ε, πολλούς ενδιαφερόμενους και προσπάθησα να ενημερώσω τους κοιόδες εισηγητής. Ε, εισηγητές. Η κυρία είναι ε, συναντήθηκε μαζί μου και με τους υπόλοιπους κοιόδες εισηγητές και είπαμε ότι δεν γίνεται να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις πριν να έχουμε εντολή από το Συμβούλιο, αλλά ελπίζω να υπάρξει εντολή γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε, μπορούν να βρεθούν λύσεις και σε ευαίσθητα θέματα όπως το άρθρο 7. Αυτή τη στιγμή αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Πιέζουμε λοιπόν, αλλά για την ώρα δεν υπάρχουν νεότερα από το Συμβούλιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που διατηρείτε την πίεση. Κρίμα. Είναι απογοητευτικό μετά από τις τεράστιες προσπάθειες που έχετε καταβάλει και εσεί και η κυρία Πιετικά είναι και η ολόκληρη επιτροπή μας να ψηφίσουμε το περασμένο μήνα για να έχουμε χρόνο να διαπραγματευτούμε. Τώρα το Συμβούλιο μας καθυστερεί. Πραγματικά πολύ απογοητευτικό αυτό για του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Είδα σύντομα τον κύριο Ταγιάννη στην, ε, στο Στρασβούργο και μας είπε ότι προσπαθούν και εκείνοι να πιέσουν για τις διαπραγματεύσεις του άρθρου 7, το οποίο προφανώς είναι το επίμαχο άρθρο. Είναι κρίμα πάντως γιατί οι καταναλωτές ε, θα είναι... Δεν θα ευνοηθούν αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις πριν τελειώσει η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Ε, φαντάζομαι θα το συζητήσετε κι εσείς με τους σκιώδεις συζητητές ε, να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία του συντομότερο δυνατόν για να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις με σαφή διαπραγμάτευση από το Κοινοβούλιο, με σαφή εντολή από το Κοινοβούλιο. Επειδή εγώ ήμουν επικεφαλής του τριμερούς διαλόγου, λείπει συνάδελφο, αλλά μπορώ να ενημερώσω εγώ. Είχαμε το πρόβλημα, συζητήσαμε το θέμα του ραδιενεργού εξοπλισμού, συζητήσαμε τα θέματα για τα οποία το Συμβούλιο εξακολουθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Δεν έχουν πλήρη εντολή ακόμη, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική η συνάντηση. Ήταν και η κυρία Ρούιλε εκεί. Και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε διάφορες λύσεις. Υπήρξε καλή ανταλλαγή απόψεων για το πώς είναι δυνατόν ε, να προχωρήσει αυτό το θέμα. Είμαι αρκετά αισιόδοξο. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Συγγνώμη κυρία Σενάλοβα που σας άφησα να περιμένετε. Να περάσουμε τώρα στην έκθεσή σας. Είστε η συντάκτρια γνωμοδότησης ε, για την γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Μεταφορών, ε, την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος e σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαρίστω να σας δώσω το λόγο και μετά να δώσω το λόγο στον κύριο Καμπ, στην κυρία Ρούλε και εγώ θα κάνω κάποια σχόλια ως σκιώδη εισηγητής. Κυρία Σενάλογα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή Μεταφορών ασχολείται με το θέμα επέκτασης των λεγόμενων e-call ηλεκτρονικών κλήσεων να υπάρξει μια διαλειτουργική ευρωπαϊκή ε, μορφή δικτύου των e-call. Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη πλειοψηφία στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πέρυσι και κατετέθησαν ορισμένες προτάσεις οι οποίες βελτιώνουν την ε, πρόταση. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην αναφορά στον αριθμό 112, ο οποίος είναι η βάση το, του συστήματος το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους ε, δωρεάν. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες για τις εκστρατείες πληροφόρησης, οι οποίες θα πρέπει να εξηγούν ε, τα πλεονεκτήματα των νέων αυτών συστημάτων. Οι συνάδελφος Τούν και η τροπολογία της 6 λέγουν ότι μια τέτοια εκστρατεία θα πρέπει να προηγηθεί στην ανάπτυξη του συστήματος και θα πρέπει να οργανωθεί από την συγκεκριμένη επιτροπή. Επίσης πρέπει να αναφερόμαστε στην προστασία δεδομένων που είναι ένα ε, πολύ σημαντικό θέμα γιατί ε, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το e-call δεν επιτρέπει εντοπισμό του οχήματος ε, ή καταγραφή του δρομολογίου. Συμφωνώ με αυτές τις ε, τροπολογίες, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο περαιτέρω. Επίσης, ως προς το θέμα της προστασίας ε, δεδομένων, η κυρία Τιούν προτείνει η διαχείριση της προστασίας των ε, δεδομένων να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το θέμα αυτό. Τροπολογία 4 ζητά από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν κατάλληλη χρήση μεταφοράς δεδομένων. Στην τροπολογία 12 ο ίδιος συνάδελφος ε, ζητά τα δεδομένα αυτά που θα μεταφέρονται μέσω του e-call να χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις. Μίλησα με τον κύριο Χόλτερ και συμφωνήσαμε ότι θα κατατεθεί προφορική τροπολογία. Γιατί τα δεδομένα τα οποία αντλεί κανείς από ατυχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, για προειδοποίηση ορισμένων ε, οδηγών να αποφύγουν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο που έχει γίνει ένα ατύχημα. Τροπολογίες 8 και 11 του κυρίου Φαντενκάμπ το επίπεδο ακρίβειας ε, εντοπισμού ε, του τηλεφωνήματος στο e-call από ένα ε, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, πρέπει να είναι, και, να είναι ίδιο με αυτό που γίνεται από μια συσκευή e-call. Αυτή τη στιγμή θα αρχίσει να ισχύει το σύστημα από τον Οκτώβριο του 2015. Εγώ συμφωνώ με την ίση ε, πρόσβαση στο 112 για όλους τους πολίτες. Είναι μια καθολική υπηρεσία. Είναι βέβαια ε, πέραν του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί που δυσχεραίνουν την ίση πρόσβαση που ζητούμε. Επίσης, είναι επικίνδυνο να θεωρηθεί προαπαιτούμενο η συγκεκριμένη ε, οδηγία για την ευρύτερη οδική ασφάλεια Πιστεύω όμως ότι πρέπει η διάταξη αυτή να υπάρξει τουλάχιστον σε ένα εκτιμώντας. Τα κράτη-μέλη τα οποία ζητούν η επίγουσα κλίση να είναι διαθέσιμη από όλα τα τηλέφωνα σε όλες τις χώρες ε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ελπίζω ότι ο συνάδελφος δεν θα δυσαρεστηθεί πολύ που δεν συμφωνώ με αυτή την ε, ε, τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντερκάμπ έχει το λόγο σαν σκιώδης από το ΕΛΚ. Eh, allemaal een bijzonder eh, goede morgen nog. Ik wil op de eerste plaats de rapporteur bedanken voor de doortastende aanpak. Eh, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ δραστήρια γύρω από τα θέματα αυτά. Ήρθε σε επαφή με τους κοιόδης εισηγητές το σύστημα αυτών των κλήσεων ε, ε, το διαλειτουργικό δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αν δεν εξηγηθεί σωστά. Έχουν κατατεθεί και δύο τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται ε, στην λειτουργία των συστημάτων 1 και 2 και όχι γενικότερα και αποκλειστικά με το θέμα των ηλεκτρονικών κοινών κλήσεων. Ε, το σύστημα 1 και 2 δεν υπάρχει σε όλες ε, βέβαια τις χώρες ή και αν υπάρχει υπάρχει με διαφορετικό τρόπο. Το σύστημα αυτό καλύπτεται από την οδηγία την λεγόμενη καθολικών υπηρεσιών ωφέλειας Με αυτήν λοιπόν την γνωμοδότηση για τις ηλεκτρονικές κλήσεις μπορούμε να καταλήξουμε με τις ρυθμίσεις των συστημάτων 1 και 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάσταση αυτή δεν την βρίσκει πολύ ικανοποιητική και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε. Σαν παράδειγμα στον τομέα της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων. Η τροπολογία αναφέρεται σε ε, κατεπίγουσες καταστάσεις, emergency situations. Και γι' αυτό ακριβώς αναζητάτε η αποτελεσματικότητα του συστήματος και γι' αυτό ε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα μπορούσα να ψηφίσω και σήμερα το πρωί που λέει ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ. και από δικής μου πλευράς θα συμφωνήσω με την άποψη των εισηγητρίας και δεν θα πρέπει να υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία διών. Για το θέμα του 112, ξέρετε ότι θα οργανώσουμε σήμερα το απόγευμα μια, μια ακρόαση ε, για την αγορά των ηλεκτρονικών ε, τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Και εγώ φυσικά που είμαι υπέρ της οδηγίας ε, για τις λεγόμενες καθολικού τύπου υπηρεσίες δεν θα ήμουν κατά των απαιτούμενων ρυθμίσεων. Έχουμε μια δυνατότητα λοιπόν να το συζητήσουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης η οποία έχει ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι μπορώ να διαπιστώσω με ευχαρίστηση ότι εμείς ε, λάβαμε υπόψη και τη γνωμοδότηση ε, του ελεγκτή ε, σεβασμού που ασχολείται με τα θέματα του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κύριος Ντεπρέ. Όχι, η κυρία Ντεπρέ, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής μας θα ήθελε το λόγο, αλλιώς θα δώσω απευθείας το λόγο στην κυρία Ντεπρέ. Θα σας ακούσουμε με προσοχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. από τότε που ξεκινήσαμε ε, να εξετάζουμε το θέμα αυτό, γενικότερα συμφωνούμε αν μεταξύ μας Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Ε, είναι θετικές οι περισσότερες από τις τροπολογίες οι οποίες είχε κατατεθεί και η συμβιβαστική τροπολογία την οποία προτείνει η κυρία Σενάλοβα για την εκστρατεία πληροφόρησης, ε, η τροπολογία επίσης για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μας βρίσκει σύμφωνος για την τροπολογία 10, ε, θα συμφωνήσουμε μαζί σας, δεν θα την υποστηρίξουμε. Αυτό έχει αρκετά μεγάλη σημασία για μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αν αφαιρεθεί η υποχρέωση της ανάπτυξης του συστήματος, ε, θα, στην ουσία θα ακυρωθεί η ίδια η έκθεση και η δική σας και η πρόταση η δική μας και γι' αυτό την 10 δεν θα τη στηρίξουμε. Λίγα λόγια για την τροπολογία υπαρίθμου 8 και την τροπολογία υπαρίθμου 11. Για τις δύο αυτές τροπολογίες νομίζω ότι σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοούμε πλήρως ε, τους στόχους αυτών των τροπολογιών μόνον οι ε, πολίτες οι οποίοι έχουν μέσα χρήσης ε, των e ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες εντοπισμού DNSS. Τώρα δεν θα εμείνουμε σε θέματα όπως η νομική βάση και θα επανέλθω σε θέματα περισσότερο τεχνικά. Αυτό το οποίο από πλευράς μας αποτελεί ε, έναν φόβο είναι ότι λόγω ε, μπαταρίας, κατανάλωσης της μπαταρίας, ε, ο κόσμος πολλές φορές οι χρήστες σβήνουν την, την, τη διαδικασία, την τεχνολογία που έχει το μηχάνημά τους για τον γεωγραφικό εντοπισμό, το GNSS. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα είναι το τι γίνεται με την ανάληψη ευθύνης ε, όταν είναι κανείς σε ένα κτίριο κλειστό όπως μια σύραγγα ή ένα κτίριο χαμηλά και δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν ξέρω, μήπως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί στο συγκεκριμένο θέμα και δεν ξέρω αν μπορούμε να το στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο, ο κύριος Χάμπορ. Να επιβεβαιώσω ότι εμείς θα ψηφίσουμε την συγκεκριμένη πρόταση αύριο μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών. Η κυρία Σενάλοβα μπορεί να κλείσει τη συζήτηση εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ ε, πολύ. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Με χαρά θα περιμένω την αυριανή ψηφοφορία και αγωνία. Να σας καλέσω άλλωστε και στην αυριανή, αυριανή μας ακρόαση ε, σε σχέση με το e-call. Να σας προσκαλέσω. θα είναι μια ακρόαση στην οποία θα παραστεί και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Θα είναι ο, ο συντονιστής επίσης του πιλωτικού προγράμματος, ε, θα είναι μεταξύ των ε, ομιλητών. Εξετάζει το επίπεδο ετοιμότητας των κρατών μελών ε, σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα του διασυνοριακού, της διασυνοριακής τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα του e-call. Οπότε θα ήθελα να σα καλέσω σε αυτήν την ακρόαση. Ναι βεβαίω λέει ο πρόεδρο και εγώ να σα ενθαρρύνω είτε να παραστείτε είτε να την παρακολουθήσετε μέσω ίντερνετ 11 η ώρα αύριο μετά τι ψηφοφορίε. Θα έχουμε χρόνο, μία ώρα, από τις 11 ως τις 12 για την ακρόαση αυτή, γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά και καλό είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση που καλύτερα είναι να λυθούν. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή και γι' αυτό ακριβώς ε, ε, την δουλειά της ε, κυρίας Σενάλοβα τη χωρίσαμε στα δύο για να μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε για τη μία από τις δύο και την άλλη που θα την εξετάσουμε αύριο θα την ψηφίσουμε το Δεκέμβριο για να ευθυγραμμιστούμε και με το πρόγραμμα της Επιτροπής Μεταφορών. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να σας πω είναι ότι συμφωνήσαμε με τη βοήθεια της κυρίας ε, Σενάλοβα, με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η οποία συμφωνία αφορά κάποιες πτυχές ε, της προστασίας των πολιτών. Ε, υποθέτω ότι θα μας στείλουν και εκείνη μια γρήγορη απάντηση. Φαντάζομαι ότι ό,τι έχουμε συμπεριλάβει στις αιτιολογικές σκέψεις θα καλύψει κάποιες από τις ανησυχίες, του, από τις ανησυχίες της Επιτροπής αυτής. Το είπε και η κυρία Σενάλοβα. Τα δεδομένα από το σύστημα ECOL αφορούν το όχημα, δεν είναι υποχρεωτικά προσωπικά ε, δεδομένα. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται και αυτό. Αφορά τα στοιχεία του οχήματο. Το σύστημα θα λειτουργήσει σε περίπτωση ατυχήματος ε, ε, και η κλίση θα γίνει από το όχημά του. Ο Άξελ Βος θα είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα γιατί ο κύριος Λόκεγκαρτ που αντικαθιστά τον κύριο Σμιτ είναι εδώ και νομίζω ότι και όλοι οι σκιώδες είναι εδώ. Οπότε είναι εδώ η κυρία Ράπτη, η κυρία Ρούλε και εγώ και μπορούμε να αρχίσουμε για τη γνωμοδότηση, για τη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Οικονομικών ε, τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάση των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ και ο κύριος Κιούπικ από την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ε, κάνει και εκείνος τις παρατηρήσεις του. Κύριε Λόκιγκαρντ, να σας δώσω το λόγο για να μας πείτε ποια είναι η άποψη του εισηγητή, του κυρίου Σμιτ, για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Όλες σας χαιρετά. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα γιατί είναι στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Άντις. Οι Σκιώδης ε, θεωρεί όλε ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στις τροπολογίες στις συμβιβαστικές 1 και 3 βασίζονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, ομαδικές ή συλλογικές αποζημιώσεις και για τις επιπλέον δαπάνες θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα opt-in εθελοντικής συμμετοχής. Συμφωνεί ο κύριος Σμιτ ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία ε, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί από το α μέχρι το σ αγγλικό θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν πάρα πολλές ε, διάφορες σχετικά με το επιπλέον κόστος. Εκτός από το θέμα της έλλειψης ε, πληροφοριών, η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη. 17 Δεκεμβρίου θα γίνει κανονικά η ψηφοφορία και όταν γυρίσει από την Άντις Όλε θα σας κάνει πιο συγκεκριμένες συμβιβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Λόκεργαρντ. Δεν ξέρω, ισχυώδεις ε, έχουν το λόγο ο κύριος Σβάμπ. Πρώτος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Λόκεργαρντ πάρα πολύ συνοπτικά ε, συγκέντρωσε την προσοχή μας στα ε, βασικά σημεία ε, τα οποία δημιουργούν πιθανά προβλήματα στην έκθεση του κυρίου, του κυρίου Σμιτ. Συγγνώμη. Ζήτησε να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι αλήθεια ότι τον ε, ε, Ιανουάριο θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ξέρετε ότι αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έχει αμφισβητηθεί και η νομική βάση από ό,τι φαίνεται σχετικά με την συγκεκριμένη πρόταση και από ό,τι φαίνεται επίσης και στο Συμβούλιο δεν υπάρχει ε, η απαιτούμενη ομοφωνία ε, και ε, το χρονοδιάγραμμα φαίνεται προβληματικό. Λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε την απόφαση στην φάση την οποία χρονική εμείς περιμέναμε να το κάνουμε αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τον κύριο Σμίτ όπως μας εξήγησε και ο κύριος Λόκεργαρντ. Για το σύστημα opt-in αυτό είναι μια καλή υπόθεση αλλά νομίζω ότι όλα τα θέματα που αφορούν τις συλλογικέ αποζημιώσεις θα πρέπει να καλυφθούν και από τη σύσταση του Συμβουλίου μας το επιβεβαίωσε και ο Επίτροπος. Κάποια σημαντικά στοιχεία της συλλογικής αποζημίωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας, αν και στα πλαίσια της συγκεκριμένης οδηγίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι το ευρωπαϊκό μοντέλο θα πρέπει να ακολουθήσει τη λογική του opt Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχω κατανοήσει βέβαια πλήρως. Μετά από αυτά τα οποία μας είπε θα πρέπει να σταθούμε προσεκτικά στο 2-2 και στο 13-2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι ε, απόψεις τις οποίες είχαμε από πλευράς των δικαστικών κύκλων μας επιβεβαιώνουν ότι αυτός ο οποίος ζητά να αποζημιωθεί δεν έχει την βεβαιότητα ότι θα το κάνει αυτό και επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση οι ζημίες αυτές να θίξουν και τον λεγόμενο έμεσο αγοραστή. Αν ζητήσει αποζημίωση λοιπόν και ο έμεσος αγοραστής σύμφωνα με το 13.2 φοβάμαι ότι η κατάσταση περιπλέκεται με τέτοιο τρόπο και ε, θα πρέπει ε, ο πρώτος συμβαλόμενος να πληρώσει δύο φορές ε, την αποζημίωση. Αυτό είναι μία θα έλεγα τιμωρητική διαδικασία την οποία δεν θα επιθυμούσαμε να λειτουργήσει στην Ευρώπη. Αλλά δεν έχω πείσει ακόμα το κύριο Σμιτ, είναι υποσυζήτηση το θέμα. Για τα υπόλοιπα θέματα στα οποία στέκεται ο κύριος Σμιτ στα πλαίσια των συμβιβαστικών τροπολογιών του, εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει ε, επιτρέψει κάποια έγγραφα σε μόνιμη βάση και άπαξ να είναι ε, συμβουλεύσιμα, να μπορεί κανείς να ανταχρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει μια τέτοια βεβαιότητα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναζητήσουμε ε, μια συμβιβαστική λύση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Σμιτ διαφωνεί με την πρότασή μου η οποία βασίζεται στην κάθε φορά απόφαση του δικαστηρίου. Θα πρέπει να λαμβάνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση υπόψη διάφορα στοιχεία όπως ακριβώς και αυτή η ελεγχόμενη μορφή επίοικιας αν θέλετε η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση μη ύπαρξης δόλου. Λόγω λοιπόν των συγκεκριμένων προτάσεων του κυρίου Σμιτ έχουμε βρεθεί στην, στην κατάσταση στην οποία είμαστε τώρα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το δικό της κείμενο ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα θα ξεπεραστούν, αλλά αν η λύση την οποία προτείνουμε καταστήσει την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων πιο δύσκολη και αν πράγματι θέλουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου δεν θα πρέπει να ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου σε άλλα θέματα και να περιπλέξουμε τις εργασίες του Συμβουλίου. Συνεπώς, οι συμβιβαστικές προτάσεις του κ. Σμιτ δεν είναι ακόμα αποδεκτές. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Σουάμπ. Αναφέρομαι ειδικότερα στον κύριο Σουάμπ γιατί ε, χάρηκα που τον είδα, είχα καιρό να τον δω, αλλά με αυτά που είπε με στεναχώρεσε. Ε, και με στεναχώρεσε για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι ο κύριος Σμιτ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτή την υπόθεση των συλλογικών προσφυγών. Ε, η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή Όντως, είναι μια πολύ ε, συμπαθής πρόταση. Όμως, λείπει για μια ακόμη φορά το στοιχείο εκείνο που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Το στοιχείο εκείνο που θα δείξει ότι η Επιτροπή είναι επιτέλους έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα και να είναι στο πλάι των Ευρωπαίων πολιτών. Τι λείπει από την πρόταση της Επιτροπής? Η υποχρεωτικότητα. Το να είναι υποχρεωτικό το collective redress. Πάμε τώρα σημείο προς σημείο. Το πρώτο και βασικό σημείο, θέλω να το επαναλάβω, είναι θερμές ευχαριστίες προς τον κύριο Σμιτ. Διότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά, επέδειξε συνεργατικό πνεύμα, είχε, ε, έκανε πραγματικά μια ειλικρινή προσπάθεια να βρει συνένεση και να βρει αυτό που λέμε τη χρυσή τομή. Ε, άρα η στάση του είναι όχι μόνο καθοριστική αλλά χρησιμοποιώ και τη λέξη καταλυτική για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Όταν βέβαια ακούω εγώ για νομικές βάσεις, ε, για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν κάπου μπαίνει και η Επιτροπή γιουρί στη μέση, αμέσως αρχίζω και φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πάμε για αναβολή και ξανά αναβολή και για μια ακόμη φορά αυτό το πολύ ταλαιπωρημένο θέμα των collective redress πάμε να το σπρώξουμε προς τα πίσω. Ο κύριος Σουάπ κατέληξε ε, κάνοντας ουσιαστικά ε, έναν έμεσο, πολύ λεπτό και διπλωματικά διατυπωμένο εκβιασμό. Είπε, εάν θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση των collective redress σε αυτή την ομοθετική περίοδο, να μην ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου. Πρώτον, θέλουμε όλοι και είναι καλό και πρέπει για το καλό των ευρωπαίων πολιτών να τελειώσουμε με τις συλλογικές προσφυγές σε αυτή την νομοθετική περίοδο. συμφωνούμε. εκείνο όμως που υπόθηκε για τους ασκούς του αιώλου αυτό με φόβησε. θεωρούμε ασκό του αιώλου το να είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τον ευρωπαίο καταναλωτή. εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ασκός του αιώλου θεωρώ ότι είναι πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας κοινωνικής ευρώπης για την οποία όλοι μιλάμε και για την οποία όλοι υποτίθεται ότι παλεύουμε ιδιαίτερα πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Ε, πηγαίνω τώρα στις συμβιβαστικές. Οι πρώτες δύο συμβιβαστικές έχουν την απόλυτη υποστήριξή μας ο κύριος Σμιτ έκανε και εδώ πολύ καλή δουλειά. Στις συμβιβαστικές 3 και 4 έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε όλο τον καιρό να το χειριστούμε. Και αυτό γιατί η πρόταση η δική μας είναι να επεκτείνουμε το μαχητό τεκμήριο βλάβης λόγω παραβίασης του δικαίου του ανταγωνισμού, όχι μόνον στα καρτέλς. Κλείνοντας, ε, θέλω για μια ακόμη φορά να πω ότι συμφωνώ και στηρίζω τις βελτιώσεις και τις αποτελεσματικές λύσεις που προτείνει ο κύριος Σμιτ και ε, στηρίζω και το θέμα του χρονοδιαγράμματος, το γεγονός δηλαδή ότι πάμε πίσω την ψηφοφορία. Αλλά εδώ θέλω να κάνω και δύο επισημάνσεις, αν θέλετε δύο παρακλήσεις. Η μία παράκληση είναι προς όλους μας. Τους ευρωβουλευτές, την Κομισιόν, τις υπηρεσίες, τις γραμματείες, τους πάντες εν πάση περιπτώσει όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τελειώσουμε, να ψηφίσουμε για το θέμα των συλλογικών προσφυγών σε αυτή την ομοθετική περίοδο. Η δεύτερη παράκληση απευθύνεται στο ΕΠΠ και προσωπικά στο φίλο μου, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη δουλειά του, τον κύριο Σουάμπ. Είναι εισηγητής για το θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών. Είναι εδώ ο σκιώδης Αυτό το θέμα το έχει πάρει αγκαλιά ο κύριο Σουάμπ. Τον παρακαλώ πάρα πολύ να μην το σφίξει, μην σφίξει πολύ αυτή την αγκαλιά γιατί θα το πνίξει το θέμα. Και αν το πνίξει θα είναι σαν να πνίγουμε και να στερούμε το οξυγόνο από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. η κυρία Ρούλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σμιτ για την εξαιρετική δουλειά και υποστηρίζουμε όλες τις προτάσεις τροπολογιών τις οποίες έχει καταθέσει. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πάρω και εγώ το λόγο σαν σκιώδης από πλευράς της δικής μου πολιτική ομάδας. Έχουμε κάποιες ανησυχίες με κάποιες από τις συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες βρίσκονται κατ' εμέ σε προπαρασκευαστική ε, φάση θα έλεγα. Ξέρετε, είπα στην αρχή της συνεδρίασης ότι αναβλήθηκε η ψηφοφορία γιατί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θα καθυστερήσει. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο για να εξετάσουμε τις συμβιβαστικές. Το βασικό μας πρόβλημα και εδώ θα το σχολιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει σχέση με το ότι για να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε τους καταναλωτές να ζητήσουν αποζημίωση για τη συμπεριφορά των καρτέλ, Πολλές φορές ο, ο καταναλωτής ε, δεν θίγεται άμεσα με την έννοια ότι αγοράζει ένα προϊόν μέσω ενός άλλου προμηθευτή, μέσω ενός λιανικού εμπόρου σαν παράδειγμα. Δημιουργείται μια αλυσίδα θα έλεγα στις ζημίες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πώς μπορεί η υπεράσπιση του καταναλωτή να ωφεληθεί από τη διαδικασία της απόδοσης ευθύνης στην αλυσίδα η οποία έχει προηγηθεί. Έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες για να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες μέχρι τώρα δεν έχουν αντιμετωπίσει το θέμα και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθεί σε αυτό γιατί την απασχολεί και την ίδια. Ε, κάποιος άλλος θα ήθελε να κάνει κάποια επιπλέον σχόλια. Όχι από τα μέλη. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει τη δική του άποψη. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη γενική υποστήριξη της Επιτροπής σας ε, για την ε, πρότασή μας. Επίσης χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που φαίνεστε αποφασισμένοι να προσπαθήσετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν ε, τις ευρωεκλογές. Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα θέματα, είναι γεγονός ότι... Το πέρασμα τη ευθύνη ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίω. Ε, είναι σημαντικό γιατί μερικέ φορές από την αλυσίδα φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδα και στον τελικό καταναλωτή. Και είναι δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό γιατί είναι πέρα από τη διαδικασία της παράβασης και επίση, μερικέ φορές δεν υπάρχει και άμεση πρόσβαση στα ε, έγγραφα που χρειάζονται για να αποδειχθεί αυτό που τελικά έχει καταλήξει να είναι στο δικό τους επίπεδο Υπάρχει λοιπόν ένα, μια λάφρυνση του άχθους αποδείξεως για τους έμεσους ε, ε, αγοραστές και ίσως ο κύριος Σμιτ μπορεί να δουλέψει επί της ε, κατάλληλης προειδοποίησης για να γίνει και αυτό σεβαστό. Οι κανόνες της μετάβασης ευθύνης είναι σημαντικοί γιατί η αποζημίωση πρέπει να πηγαίνει στο επίπεδο όπου υπήρξε η βλάβη. Δηλαδή, αν το καρτέλ ε, είχε δημιουργήσει μία βλάβη σε διάφορα επίπεδα, δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτός ε, που είναι υπεύθυνο να ε, ξεφύγει, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι ο εναγόμενος θα μπορούσε να πει ότι η ευθύνη μετακυλίστηκε σε επόμενο επίπεδο. Πρέπει όμως αυτή την περίπτωση να υπάρχει κάποιο είδους αποζημίωση τουλάχιστον κάποιο, κάποιο βάρος απόδειξης και σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει περαιτέρω αν χρειάζεται όσον αφορά τώρα τις ε, συλλογικές αποζημιώσεις. Πρέπει να πω ότι αυτό το θέμα το συζητούμε εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο και στο τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ακολούθησε την άποψη του Κοινοβουλίου του 2011 για το θέμα αυτό, δηλαδή οριζόντια προσέγγιση που καλύπτει όχι μόνο το δίκαιο του ανταγωνιστού μου, αλλά και του καταναλωτικού δικαίου και άλλους τομείς παραβίασης ε, ε, του δικαίου. Αυτό κάναμε Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και μία πρόταση για συλλογικές αποζημιώσεις που, ζητούν, που ζητά από τα κράτη-μέλη εντός δύο ετών να έχουν διαδικασίες συλλογικών αποζημιώσεων. Βέβαια είναι μία σύσταση, οπότε δεν είναι δεσμευτική, αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής συζήτησης που είχαμε. Και ένας από τους λόγους ήταν ότι μία από τις διαφορές, ε, ε ότι κάποιες από τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι τεράστιες αυτή τη στιγμή, ε, ξέρετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εισαγάγει ε, τεράστιες αλλαγές στο δίκαιο ανταγωνισμού ε, και ξέρετε ότι και στη Γαλλία και στο Συμβούλιο και στο Βέλγιο τα κοινοβούλια συζητούν το θέμα των συλλογικών αποζημιώσεων. Οπότε, επειδή είμαι και υπάλληλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υποστηρίξω τα πεπραγμένα τη όταν ακολούθησε την οριζόντια προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ε, ο, αν, αν για τον τελικό χρήστη δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογική προσφυγής, τότε ο καταναλωτή στο τέλος δεν έχει και τίποτε στα χέρια του. Θέλουμε λοιπόν από τη μία να υπάρχει μεγαλύτερη αποζημίωση, ε, είναι, καλύπτεται από τη συγκεκριμένη πρόταση, θα καλύψει όλες τις προσφυγές, ακόμη και τις συλλογικέ και μετά το επόμενο βήμα είναι η σύσταση για τις συλλογικέ προσφυγές αυτές καθεαυτές και αυτό βέβαια θα το δούμε σε επόμενο στάδιο αν δούμε ότι σε δύο χρόνια τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακολουθήσει τη σύσταση αυτή. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως ε, να συζητήσει περαιτέρω κάτι ακόμη ο κύριος Φαμπ αμφιβάλλει για την απόλυτη ε, για τις δηλώσεις ανάληψης ευθύνης ε, και κατά πόσο ευθυγραμμίζονται ε, με την νομολογία. Όμως, αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο, μπορούμε να ακολουθήσουμε την νομολογία. Τότε το δικαστήριο θα έλεγε, ο δικαστής είναι αυτός που θα αποφασίσει τα πράγματα κατά περίπτωση. Θα αποφασίσει κατά περίπτωση. Ένα δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι και εκείνο έτσι ερμηνεύει την ομολογία και ε, η στάθμιση του ε, δημοσίου συμφέροντος ε, και του ιδιωτικού συμφέροντος ε, αποζημίωσης είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη με έναν λογικό τρόπο. Είναι κάτι βεβαίω το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος ε, Χάρμπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντησή σας. Κύριε Λόκεγκαρντ, να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κύριε Λόκεγκαρντ. Ναι, βεβαίως, όλα αυτά τα σχόλια θα τα μεταφέρω στον Όλε. Βεβαίως ε, θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σχόλια στις ε, επόμενες συζητήσεις. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο ότι στις 15 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε ο κύριος Σμιτ θα έχει τη δυνατότητα ως τότε να, να ανταποκριθεί σε κάποιες από τις ανησυχίες ε, που ακούστηκαν για τις συμβαστικές τροπολογίες πριν την ψηφοφορία της 17ης Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Λοιπόν, για όσους δεν ήσασταν εδώ νωρίτερα, να πω ότι το επόμενο θέμα θα είναι η έκθεση του κυρίου Λόκιγκαρντ για το Solvit. Έχουμε πάει μια φορά πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό δεν είναι σημαντικό, και είναι δεν, είναι, δεν είναι εδώ και είναι σημαντικό να είναι εδώ για να, ακούσετε αυτά, να ακούσει αυτά που έχει να πει ο κύριος Λόκεγκαρτ. Όμως περισσότεροι σκιώδεις εισηγητές είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Μπέλα είναι εδώ. Καλημέρα σας. Η κυρία Χάντζλικ δεν είναι εδώ. Κύριε Σφάπ, την αντικαθιστάτε. Μάλιστα, και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για τη δική μου ομάδα και η κυρία Ρούλε φαντάζομαι το ίδιο. Οπότε, προτείνω να διακόψουμε λίγο μέχρι να έρθει η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί φαντάζομαι κύριε Λόκεγκαρτ θέλετε να είναι εδώ η Επιτροπή, να ακούσει τι έχετε να πείτε για το σχέδιο έκθεσής σας που είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε λοιπόν να βγείτε για λίγο, για ένα καφεδάκι, παρακαλώ να γυρίσετε το συντομότερο δυνατόν, γιατί μόλις έρθει εκπρόσωπος κυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξαναρχίσουμε. Uh, uh, λοιπόν, να ξαναξεκινήσουμε επειδή νομίζω όλοι οι επικεφαλής είναι εδώ η κυρία Χάνσλικ μόλις έφτασε ως σκιώδης συγγήτρια εκείνη. Λοιπόν, επίσης καλωσορίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρίσταται. Καθώς κάθονται τα μέλη να πω ότι αυτό είναι ένα νέο newsletter ενημερωτικό δελτίο που μόλις ε, διατύπωθηκε και διανεμήθηκε. Και στο διαδίκτυο όσοι μας παρακολουθείτε μπορείτε αν ζητήσετε από την ιστοσελίδα να το αποκτήσετε και να το έχετε στη διάθεσή σας. Θα δείτε εξέχουσες προσωπικότητες στην πρώτη σελίδα και της αποστολής ε, στην Κίνα. Είναι και ο κύριος Σβάμπ και η κυρία Χάνσλικ. Οποιοςδήποτε θέλει να τα διαβάσει αυτά εμπεριέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Λοιπόν περνάμε τώρα και θα ακούσουμε από τον κύριο Λόκεγκαρντ, τον εισηγητή μας που μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του για το Solvit. Και μετά θα καλέσουμε τους σκιώδεις εισηγητές να σχολιάσουν επίσης Χάσλικ, Αμπέλα και η κυρία Ρούιλε. Άγκστρομ επίσης, εντάξει ωραία. Ένας από τους πράσινους συναδέλφους, ευχαρίστως να έχουμε και παρέμβαση και εγώ θα έχω και παρέμβαση από την ομάδα μας και από την κυρία Γκρόβινς που είναι φίλη της Επιτροπής μας και παρίσταται Ανούσκα Γένσενς επίσης που εκπροσωπεί την κυρία Γκρόμπεν η κυρία αυτή θα σχολιάσει την έκθεση από πλευρά σας. Κύριε Λόκεγκαρτ σας δίνω αμέσω τον λόγο. Παρακαλώ. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συγχαρητήρια με την πολύ επιτυχή επίσκεψη στην Κίνα Ίσως θα μπορούσα και εγώ να είχα συμμετάσχει ευχαρίστως, αλλά μια άλλη φορά έστω. Εντάξει. Τώρα, με τους συναδέλφους, περνώντας σε αυτό το θέμα του Solvit, να πω το εξή. Είχαμε συζητήσεις και έχω την εντύπωση του γνωστού ήδη, déjà vu. Θυμάμαι και την αποστολή στη Στοκχόλμη πριν από τέσσερα χρόνια. Ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι. Συζητήσαμε πολύ για το Solvit με τις Σουηδικές αρχές τότε και δεν μπορούσα να διαφύγω τη συνέστηση ότι είχα ακούσει ακριβώς τα ίδια πράγματα στο παρελθόν, τις ίδιες ακριβώς συζητήσεις, με τα ίδια αριθμητικά μεγέθη και στοιχεία, όπως και πριν από τέσσερα χρόνια τότε με αυτά τα οποία λέγαμε τώρα. Καλό αυτό, υπάρχει όμως χώρος για, για βελτιώσεις εδώ, εντάξει. Αυτό που θα ήθελα να σας πω τώρα είναι ότι υπάρχει κάποια απογοήτευση από πλευράς μου, σημειώνοντας ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το Solvit, τα ίδια όπως αντιμετωπίζαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Και αυτό είναι η εκκίνηση, η αφετηρία για μένα σε αυτή τη συζήτηση. Όπως τόνισα στην έκθεσή μου, θεωρώ ότι ίσως τώρα πλέον ήρθε η χρονική στιγμή να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Solvit 2.0. 2,0. Αυτό θα σήμαινε επικέντρωση ισχυρή στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουμε πιο περίπλοκες υποθέσεις που σχετίζονται με τις εταιρείε και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουμε παράλογα ή προβλήματα όπου υπάρχει αντίφαση εθνικών διατάξεων με την κοινοτική νομοθεσία. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα πολυσχηδώς το Solvit. Πρέπει τα κέντρα να χρηματοδοτούνται καλύτερα. Τα στελέχη πρέπει να έχουν καλύτερη γνώση των, της νομολογίας το να ονοματίζουμε και να κατονομάζουμε με άλλα λόγια τους υπεύθυνου ε, ώστε να υφίστανται την ε, κατεσχήνη είναι κάτι σημαντικό. Βήματα και διαβήματα πρέπει να αναλυθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι τις πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα τις αναλαμβάνουν τα κέντρα του Solvit. Στενότερη εμπλοκή των όσων ετούνται στις διαδικασίες ε, των προσφευγόντων και ίσω και σε σχέση και με την Επιτροπή, αυτό είναι το πιο ίσω σημαντικό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα έπρεπε να δημιουργήσει συγκρίσιμα στοιχεία και βέλτιστε προδιαγραφέ ω ορόσημα, ώστε να μπορούν να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Αυτό με οδηγεί στην τελευταία μου παρέμβαση, που είναι και η πιο επίμαχη, πιστεύω. Θεωρώ, αν αυτοί οι στόχοι δεν επιτευχθούν, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο, α το πω έτσι, ανοίξουμε την πύλη, την θύρα, να δούμε μήπως θα αντικατασταθεί η άτυπη διαδικασία με νομοθετική διαδικασία. Το λέω αυτό ελεύθερα και ενσυνείδητα ε, κάνοντας χρήση ε, της ελευθερίας πρότασης, υποβολής πρότασης να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε τα κέντρα του Solvit να βρίσκονται ακριβώς στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης για την ενιαία εσωτερική αγορά για το 2020 ως χρονορίζοντα, πρέπει πιστεύω να συνειδητοποιήσουμε τι συνεπάγεται να, και τι πρέπει να γίνει για να φτάσουμε εκεί. Όχι να συνεχίσουμε με λόγια και συζητήσεις συζητώντας και λέγοντας ότι τα κέντρα Solvit είναι ωραία και καλά, αλλά να δούμε τι πρέπει να γίνει για να επιτύχουμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο και γι' αυτό λέω σε σχέση με το άρθρο 25, το εδάφιο 25 στην έκθεσή μου, όπου πραγματικά αναφέρω αυτό το θέμα. Και φυσικά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, τις θέσεις σας για αυτό το 25 να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασης άτυπης διαδικασίας με νομοθετική πράξη. Να τα συζητήσουμε αυτά ανοιχτά, με ανοιχτό πνεύμα. Να καταφέρουμε η πραγματική συζήτηση να ξεκινήσει πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε το Solvit να περάσει και να λειτουργήσει στο επόμενο επίπεδο όπως χρειάζεται. Ολοκληρώνω εδώ. Ευχαριστώ. Thank um, Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Έχετε δίκιο θα έλεγα σίγουρα να εξετάζετε πώς μπορούν να προαθούν τα πράγματα με κάποιο τρόπο. Σας ακούσουμε τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών. Ξεκινάμε με σας κύριε Χάνσλικ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω τον εισηγητή και να τον συγχαρώ για μια εξαιρετική δουλειά. Έχω την αίσθηση του ντεζαβί βέβαια, γιατί πράγματι αυτά παραπέμπουν στις προηγούμενες συζητήσεις τις οποίες είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας είναι μια καλή γνωμοδότηση και με την οποία συμφωνώ. Το Solvit ίσως να μην είναι μια απόλυτα πετυχημένη διαδικασία. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι το δυναμικό το οποίο ενυπάρχει στο σύστημα δεν έχει γίνει πλήρως αντικείμενο εκμετάλλευσης και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ε, βελτίωσης. Χαίρομαι που ο εισηγητής συγκεντρώνει την προσοχή του σε θέματα πρόσβασης και σε θέματα ενημέρωσης για περισσότερη πρόσβαση. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί η ενημέρωση των ε, Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει τα μάλα στην βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτό το οποίο έχει επίσης σημασία είναι να είναι σωστά εκπαιδευμένο το ανθρώπινο δυναμικό. Μόνο σωστά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Solvit θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν πλήρως και ταυτόχρονα να έρθουν αρρωγοί στους πολίτες και τους επιχειρηματίες γενικά. Το Solvit έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα μέσο το οποίο θα περιορίσει τις καταχρήσεις οι οποίες γίνονται και των δικαστικών διαδικασιών. Ίσως να υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες, κάποιες πλευρές οι οποίες ε, βιάζονται μερικές φορές να υποβάλουν ορισμένες διαδικασίες σε δικαστική εξέταση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε μια πρώτη τουλάχιστον φάση, το Solvit είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί χρήσιμο. Απαιτείται για να γίνει όμως αυτό μια σωστή χρήση των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχει το σύστημα. Οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι το Solvit είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την ανείχνευση των μη ε, κανονικών διαδικασιών στα πλαίσια της εφαρμογής του κοινοτικού νόμου. Χαίρομαι που ο εισηγητής δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε αυτό. Η εφαρμογή του κοινοτικού νόμου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ε, περαιτέρω διατήρηση των εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το Solvit είναι εξαιρετικό μέσο και για την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντοπίζει ταχύτατα τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς, τα οποία συνδέονται με τη μη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Τώρα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος μέσω μιας νομικής πλέον πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρουσιάζει το σύστημα, είναι μια δυνατότητα την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς. Το Solvit έχει μεγάλη σημασία και για τους επιχειρηματίες και δίνει την δυνατότητα να βρίσκει ανεπίσημες λύσεις σε ε, θέματα που αφορούν στους επιχειρηματίες. Λόγω όμως της έλλειψης ανθρώπινων πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και λόγω και κάποιων ε, επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κέντρα που ασχολούνται με το Solvit, ε, μερικές φορές η ανταπόκριση δεν είναι αυτή την οποία περιμένουν οι επιχειρηματίες. Είπε ο εισηγητής ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία δεν συμμετοπίσουν περίπλοκα θέματα και όμως ακριβώς εκεί βρίσκεται η χρησιμότητα του συστήματος για, το, για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για μια εξαιρετική έκθεση και θα πρέπει να συνεχίσουμε την συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό και ίσως πράγματι να εξετάσουμε και τη δυνατότητα μιας νομικά δεσμευτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάνσλε και κυρία Σαβέλα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μένα ήταν σύμπτωση, πραγματική συγκυρία ότι βρέθηκε το Solvit ε, μπροστά μου και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά με ανησυχεί και μας ανησυχεί. Δεν γνωρίζουν όλοι για αυτή την υπηρεσία για το Solvit, για αυτή τη δυνατότητα. Βλέπετε πόσοι πρέπει να είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν για αυτές τις υπηρεσίες του Solvit. Τώρα, για τις συστάσεις ε, σε σχέση και με το πρόγραμμα δράσης. Για μένα είναι θεμελιώδες και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν ε, να, να επωφεληθούν από τα προτερήματα της ευρυνίας αγοράς. Και η στόχος πρέπει να είναι στο τέλος ότι και πολίτες και επιχειρήσεις είτε έχουν προβλήματα όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες τους, κοινωνική ασφάλεια ή οποιαδήποτε άλλα θέματα να γνωρίζουν πού πρέπει να στραφούν και να βοηθηθούν να μπορούν έτσι διασυνοριακά στις ε, δραστηριότητε, τους οι πολίτες ε, να, ε, όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους πρέπει να γίνονται σεβαστά και για την ίση μεταχείριση να μπορούν να γνωρίζουν πού να στραφούν ώστε να έχουν συμβουλή που θα τους δοθεί ή να επιληθεί το πρόβλημά τους και να διασφαλίζεται έτσι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει ενεργά να εμπλακούμε ώστε να βελτιωθεί το Solvit ώστε να είμαστε αποτελεσματικότεροι και οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι στοχεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Επίσης καλωσορίζω, χαιρετίζω το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Λόκεγκαντ. Είναι σημαντικό να εμένουμε και να επιμένουμε ότι τα κέντρα Solvit ακριβώς όταν λειτουργούν και με αυτόν τον τρόπο να έχουν τα αναγκαία στελέχη και τα κονδύλια από τα, ε, τις εθνικές αρχές τους. Και η συνεργασία μεταξύ των κέντρων Solvit θα πρέπει να επιτηρείται και να βελτιωθεί και αυτή. Αυτό που είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος ε, πρέπει να είναι ότι με τις νέες συστάσεις ο ορισμός ε, των περιπτώσεων Solvit επικαιροποιείται και αυτό δίνει μια πιο συνεπή προσέγγιση για την ερμηνεία όσων πρέπει να γίνονται από τα κέντρα αυτά του Solvit. Γι' αυτό θα πρέπει τα προβλήματα να είναι ευδιάκριτα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αποτελεσματικά. Για τον ευδιάκριτο χαρακτήρα καλωσορίζω ιδιαίτερα τα σχόλια τα οποία περιέχονται στην έκθεση για τον ευδιάκριτο χαρακτήρα και των θεμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων σε σχέση με το Solvit. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται μια ολιστική, συνολική, ευρία προσέγγιση για τα εργαλεία και τα μέσα. Όχι μόνο τα κρατημέλη πρέπει να κληθούν να εμπλέκονται σε εκστρατείε ενημέρωση, αλλά επίση είναι σημαντικό να ε, δώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξη των εθνικών ιστοσελίδων και δικτύων ώστε να μπορέσουν έτσι να συνεισφέρουν σε σχέση με τις προσπάθειες όσον αφορά σημεία επαφής και δράσης. Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε όταν πολίτες ή επιχειρήσεις έχουν ένα πρόβλημα με οποιοδήποτε ε, πλαίσιο στο, στις νέες αρμοδιότητες να μπορούν ε, να στραφούν στο σωστό σημείο για να βοηθηθούν. Φυσικά οι πολίτες ε, θα πρέπει σε σχέση με το Solvit να κάνουν χρήση αυτών των δυνατοτήτων μια και είναι στη διάθεσή Ταυτόχρονα, μια και οι ιστοσελίδες και των ε, εθνικών κέντρων ε, και βρίσκονται υπό ε, συγκρότηση, υποκατάρτιση, θα πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα πρόσβαση σε αυτά και για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να συμπληρώνει την έκθεση και θα καταθέσω τροπολογία για να γίνει αυτό. Επίση, θα ήθελα να ληφθεί υπόψη όπω προηγούμενα, μια και εισήχθη αυτό από πλευρά τη Επιτροπής Απασχόληση ΕΜΠΡ, πρέπει να δοθεί ευκαιρία στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν κέντρα Solvit στο περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό φυσικά μπορεί να συνδυαστεί με άλλα γραφεία εκπροσώπησης Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώ θα μπορέσει έτσι να λειτουργήσει αυτό στο πλαίσιο τη διοίκηση, Να δοθεί μια δυνατότητα να ε, έχουμε πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερο στους πολίτες. Να έχουμε και τα εθνικά κέντρα αλλά να μπορούμε και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ταυτόχρονα να δράσουμε και με ιστοσελίδες ε, ώστε να υπάρχει συνέργεια μεταξύ ιστοσελίδων και κέντρων. Αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει νομίζω να ληφθούν υπόψη. Βρισκόμαστε στην ορθή, στη σωστή πορεία. Πολλά μπορούν να γίνουν για τη συνεργασία εθνικών κέντρων Solvit και γι' αυτό ε, προσβλέπω στη συνεργασία για αυτό το χαρτοφυλάκιο με τον εισηγητή και τους άλλους εισηγητές και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί αυτός ο οργανισμός Solvit. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μπέλα. Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Κυρία Ρούλε. Ή ο κύριος Έγκστρομ. κυριος κυρια ρουλε Θα είμαι σύντομη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι όπως και εκείνος. Δέκα χρόνια είμαι στην Επιτροπή και το Solvit είναι διαρκές πρόβλημα. Και μόνιμο και διαρκές θέμα επίσης. Από την άλλη πλευρά να μην ξεχνάμε ότι παράλληλα με το Solvit ε, έχουμε πολλά πράγματα που αναπτύχθηκαν. ADR, ε ODR, εξοδικαστικές ε, ρυθμίσεις και συμφωνίες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που παράλληλα διεξάγονται με το Solvit και αυτό πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη αν θέλουμε να έχουμε νομοθετικές πράξεις ή άτυπες διαδικασίες. Γιατί το θέμα της αναλογίας στο Solvit με νομοθετικές πράξεις θα βρισκόταν σε αντιδιαστολή με τα μέσα ADR ODR. Πιστεύω ότι πρέπει να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Δεν έχουν αποσαφινιστεί επαρκώς πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμα, πιο περισσότερο συγκρίσιμα στοιχεία και το naming and shaming, το να ονοματίζουμε τους υπεύθυνους και τους φταίχτες είναι σημαντικό. Και προς την Επιτροπή το, ερώτηση, το ερώτημα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει τέτοια στοιχεία. Από αυτό εξαρτάται. Από το να έχουμε δηλαδή συγκρίσιμα στοιχεία ως γνώμονες, ως ε, μέτρα και σταθμά με τα οποία θα μπορούμε να μετρήσουμε και να σταθμίσουμε το τι γίνεται και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις των κέντρων Solvit. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρούλε. Για το τελευταίο σημείο που αναφέρατε, συμφωνώ απολύτως και εγώ ως κοιόδης εισηγητής και νομίζω ότι μπορούμε και να το συνδέσουμε ε, ε, με τις πληροφορίες για το Solvit. Τις πληροφορίες να τις συνδέσουμε με κάποιους από τους δείκτες για την ενιαία αγορά όπως θέλουμε για παράδειγμα την εισαγωγή της διαδικασίας του εξαμήνου. Γιατί φαίνεται ότι πρέπει να προωθήσουμε πολύ περισσότερο το Solvit, αλλά πρέπει να έχουμε και δείκτες για το πού υπάρχουν τα προβλήματα, κυρίως στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Συμφωνώ απολύτως με τον τρόπο με τον οποίο ε, χειρίζεται τα πράγματα ο κύριος Λόκεγκαρτ. Ε, πολλές φορές έχουμε συζητήσει το Solvit, έχουμε κάνει πάρα πολλές ε, εκθέσεις, έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερους πόρους για το Solvit. Πιστεύουμε όμως το δημόσιο πρόσωπο της ενιαίας αγοράς ε, σε σχέση με την πρόσβαση ε, στην αγορά παραμένει πολύ κατακαιρματισμένο και επειδή έχουμε όλο και περισσότερα προγράμματα γύρω από την ενιαία αγορά, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα, όπως για παράδειγμα τα ε, σημεία επαφής τα single contact points ε, που ενημερώνουν τον κόσμο αν θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση ή αν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ε, με τα δικαιώματά του. Υπάρχει επίσης και το δίκαιο των καταναλωτών ε, σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές γενικότερα. Επίσης φαίνεται έτσι ότι στο πακέτο των ε, εμπορευμάτων το 2005 υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να υπάρχουν σημεία επαφής ε, για τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων. Δεν είχαμε όμως ποτέ ε, καταφέρει να θέσουμε μια, ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και δεν ξέρω αν υπήρξε αποτελεσματική και ικανοποιητική εφαρμογή ε, του προγράμματος αυτού. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες σε σχέση με τη μη χρήση των, των συστημάτων αυτών και της πρόσβασης ε, στα αγαθά. Μπορεί στην επόμενη σύσταση της Επιτροπής μας να είμαστε λίγο πιο ριζοσπαστικοί σε σχέση με το ε, θέμα αυτό. Πώς είναι δυνατόν να το, προωθήσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Είναι πολύ ε, κακή η χρήση του Solvit σε σχέση με το πόσες συναλλαγές γίνονται ε, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και πολλοί κόσμος δεν ε, παραπονιέται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γιατί δεν γνωρίζει πολύ απλά το Solvit. Οπότε αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο κύριος Λόκεγκαρτ λέει λοιπόν ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πώς να προσπελάσει το Solvit και το θυμάμαι και σε προηγούμενες ε, προσπάθειές μας ε, υπήρχε μια διευκόλυνση για τους ευρωβουλευτές να υποβάλουν καταγγελίες απευθείας στο Solvit ε, όσες καταγγελίες γνωρίζαμε πάση περιπτώσει έφταναν στα αυτιά μας και ήταν πραγματικά πολύ καλό και για τους πολίτες να έχουν αυτή την επιπλέον δυνατότητα υποβολής καταγγελίας. Οπότε θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα που έχουν καταγγελιών ε, στο Solvit. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι, δεν το ξέρουν. Ε, βλέπω η κυρία Χάνσλικ και πολλοί άλλοι συμφωνούν μαζί μου. Ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε τότε εσωτερικά. Αυτό να είναι ένα νέο τμήμα της δουλειάς μας, να πρωτοστατήσουμε εμείς αυτής της προσπάθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε και το σχέδιο δράσης ε, για την προώθηση της Ευρώπης σου, Your Europe. Φαντάζομαι το κύριο Λόκεργκαρντ αναφέρεται και σε αυτό. Κάπως πάντως πρέπει να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στις ε, συστάσεις μας. Και θα πρότεινα να είναι λίγο πιο ριζοσπαστικός ο κύριος Λόκιγκαρτ, να μην φοβάται στην ε, έκθεση αυτή που ε, συντάσσει για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και το πρόβλημα αυτό της προσβασιμότητας. Χαίρομαι που η κυρία Μπέλα έθεσε το θέμα της αποκέντρωσης των σημείων επαφής ε, σε περιφερειακό επίπεδο, σε πιο αποκεντρωμένο επίπεδο. Είναι σημαντικό τμήμα αυτού του πιο συνεκτικού, μιας πιο συνεκτικής πύλης που θα, έχει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ε, ζητούν αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενιαίας αγοράς με πιο επικοδομητικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για το Solvit λοιπόν 2.0, για αυτή την εκδοχή του Solvit, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο, τον κύριο Λόκιγκαρτ και ελπίζω να λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλει κανείς άλλος ε, να ε, πάρει το λόγο πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Τι Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Κρόμπεν που δεν μπόρεσε να παραστεί. Κλήθηκε σε μια επίγουσα συνάντηση ταυτόχρονα με αυτήν εδώ σήμερα σε εσά. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για την έκθεση, για το σχέδιο έκθεσης και για την υποστήριξη από την Επιτροπή σας για το Solvit. Πολλά από τα θέματα ουσιαστικά που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης καλύπτονται από το, τις νέες συστάσεις. Εργαζόμαστε στεναρά και σκληρά με τα κράτη-μέλη ώστε τα κέντρα Solvit να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να υλοποιήσουν τα διαφορετικά στοιχεία αυτά τα οποία συνιστούμε στη σύστασή μας. Και αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να καταλήξουμε στο Solvit 2 ε, το ισχυρό σημείο του Solvit είναι ο άτυπος χαρακτήρας που έχει. Το να διασαλεύσουμε αυτόν τον ε, άτυπο χαρακτήρα θα μπορούσε να οδηγήσει στο να υπονομευθεί το σύστημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ο άτυπος αυτός χαρακτήρας κάνει τα κέντρα Solvit να είναι δυνατόν να επιλύουν προβλήματα με άτυπο χαρακτήρα. Τη στιγμή που κάτι γίνεται επίσημο και νομοθετημένο, όπως διαδικασίες παράβασης ή παραβίασης, τότε είναι τελείως διαφορετικό πλέον το παιχνίδι και οι πολίτες δεν θα επιθυμούν ενδεχόμενα να ε, καταλήξουν σε ένα άτυπο πλαίσιο επίλυσης. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το άτυπο στοιχείο του Solvit και πρέπει να διατηρηθεί πιστεύω. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι στην έκθεση τώρα βρίσκεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πλέον το Solvit για την ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους και οι ευρωβουλευτές το αναφέραν αυτό. Είναι για την ιστοσελίδα το θέμα αυτό η Ευρώπη σου, Your Europe και είναι επίσης κάτι το οποίο είναι ένα από τα κύρια ζητήματα θέλουμε, επιθυμούμε να έχουμε πολύ περισσότερους πολίτες που θα προσέρχονται στο Solvit δεν θέλουμε να γνωρίζουν απλά και μόνο το όνομα Solvit 500 ή τόσοι εκατομμύρια πολίτες, αλλά θέλουμε να εμπλακούν στον αγώνα που δίνεται, να επιληθούν προβλήματα. Και η ιστοσελίδα αυτή είναι μια μεγάλη δυνατότητα με ε, μυριάδες επισκέπτες ανά μήνα. Είναι η σωστή οδός να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι τα δικαιώματά τους για αυτή την ε, ε, ιστοσελίδα, για την ε, πύλη αυτή του διαδικτύου. Να μπορούν έτσι να προσφύγουν για να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματά τους σε σχέση με την ενιαία εσωτερική αγορά. Η διασύνδεση αυτής της ιστοπήλησης στο σελίδας ε, με τα εθνικά κέντρα και εθνικές δυνατότητες πληροφόρησης είναι και αυτό σημαντικό. Να μπορέσουν τα κέντρα αυτά να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες όταν θα αναζητούν πληροφορίες ε, στο εθνικό επίπεδο να βρίσκουν την δυνατότητα να βοηθηθούν από το Solvit και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για μας, για να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που ε, θα κάνει χρήση του Solvit και περισσότεροι πολίτες να καταλήγουν στο Solvit. Μια και έχουμε όλο και περισσότερους που καταλήγουν σε αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση, αμφίδρομη δράση, feedback και να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και το θέμα των δικτών, indicators, προβληματιζόμαστε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις, ε, την κατάσταση σε σχέση με τα σημεία αναφοράς. Να είναι ευρύτερο το πλαίσιο, να μπορούν να τονιστούν θέματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη στην ενιαία εσωτερική αγορά μέσω των περιπτώσεων που καταλήγουν στο Solvit οι δείκτες όχι μόνο να ενδεικνύουν πώς τα ίδια τα κέντρα αυτών λειτουργούν, αλλά επίσης να ενδεικνύεται πώς τα κράτη-μέλη σε ένα κράτος μέλος λειτουργούν τα πράγματα ως μέρος της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Εξετάζουμε πώς μπορούμε με το βέλτιστο τρόπο να το κάνουμε αυτό, ώστε <clears throat> την επόμενη δημοσίευση που θα έχουμε κατά τα μέσα του 2014 να καλύψουμε αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, θα ήθελα και πάλι το ξέρω αυτό ότι επανέρχεται το θέμα διαρκώς και μόνιμα και ήδη και στην έναρξη του Σόλβιτ 10 χρόνια πριν και όχι μόνο 5 χρόνια πριν το θέμα των στελεχών της στελέχωσης στο κέντρο Σόλβιτ είναι ένα πρόβλημα. Χαίρομαι που αναφέρεται στην έκθεση αυτό. Χρειάζεται πίεση σε σχέση με τα κράτη-μέλη, διαρκώς πολιτική πίεση για τη στελέχωση των κέντρων Solvit. Βλέπουμε ότι σε ε, πολλά ε, σημεία δεν ε, επαρκούν τα στελέχη είτε δεν έχουμε αρκετά στελέχη, έχουμε και κέντρα με την μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, με το μεγαλύτερο αριθμό προσφυγών περιπτώσεων, με ελάχιστα άτομα. Ένα, για παράδειγμα. Πρέπει τα στελέχη και οι δυνατότητες να παρέχονται στα κέντρα αυτά να δράσουν αποτελεσματικά. Ξέρω ότι στη συγκυρία αυτή οικονομικά, με τις περικοπές στα κράτη-μέλη δεν είναι εύκολο να ζητήσει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά είναι κέρια, κρίσιμη σημασία να επιτευχθεί αυτό. Αυτά είναι τα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω αναφέρω. Σας ευχαριστώ και πάλι για το σχέδιο έκθεσης. Και όλη η πίεση και επικοδομητικές επικρίσεις είναι όλα αυτά ευπρόσδεκτα. Είναι ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το Solvit με τέτοιες δράσεις. Ευχαριστώ. Good. Uh, ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την απαιτούμενη κατεύθυνση. Κύριε Λόκερ, για το χρονοδιάγραμμα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Με χαρά διαπιστώνω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τώρα έχει γίνει σεβαστό, υπάρχει μια κάποια συνένεση για το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με πιο ριζοσπαστικό τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα, όπως ζήτησε και ο πρόεδρος άλλωστε. Αν και μένουν συζητήσεις για το τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Θα ακολουθήσουν λοιπόν συζητήσεις ανάμεσα σε μένα και τους Σκιώδης. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που είπε κυρίως η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμίσει κανείς ότι εμείς δεν ασκούμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κάνετε μια καλή δουλειά και για αρκετά χρόνια πάνω σε αυτό. Περισσότερο η κριτική την οποία κάνουμε, στρέφεται, την οποία σκούμε, στρέφεται προς τα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη τα οποία δυστυχώς δεν κατανοούν αυτά τα οποία εμείς, εσείς δηλαδή η Επιτροπή και εμείς το Κοινοβούλιο κατανοούμε. Τουλάχιστον κάποιες χώρες μέλη δεν δείχνουν να κατανοούν. Παρατήρησα αυτό το οποίο είπατε ότι απαιτείται να ασκηθεί πολιτική πίεση προς το Συμβούλιο. Αυτό είναι και το παράδοξο το οποίο αντιμετωπίζεται. Συμφωνείτε μαζί μας στην ανάγκη ύπαρξη πολιτικής πίεσης. Το θέμα είναι όμως πώς να ασκήσει κανείς πολιτική πίεση σε ένα κράτος μέλος. Αυτό παραπέμπει στη συζήτηση για τον επίσημο δεσμευτικό ε, χαρακτήρα του Solvit. Το Solvit δουλεύει εδώ και 10 χρόνια και εξακολουθούμε να λέμε πώς μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για τη σωστή εφαρμογή των Solvit τι ακριβώς ε, χρειάζεται να κάνουμε. Ίσως το καρότο να μην αρκεί, ίσως χρειάζεται και το μαστίγιο. Απαιτείται λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι ε, πολιτικά ανησυχητική. Το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι πολύ διαφορετικό και ίσως διαφορετική να είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λέγω αυτό γιατί αν πράγματι θέλουμε να πετύχουμε με το Solvit θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους τρόπους οι οποίοι να αντιμετωπίζουν κάποιες πολιτικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη εφόσον πράγματι εμένουμε στη στρατηγική του 2020 και στην στρατηγική για την ανάπτυξη. Μιλήσατε για implosion στα αγγλικά. Αν τυχόν χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μέσα και πράγματι προχωρήσουμε στην συζήτηση για νομικά δεσμευτικά κείμενα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτή την εσωτερική έκρηξη, τι ακριβώς σημαίνει, ποιο είναι αυτό το κακό σενάριο το οποίο έχετε στο νου σας. Θα ήθελα, ίσως όχι τώρα, αλλά από εδώ και πέρα στις συζητήσεις να μας εξηγήσετε τι έννοια προσδίδεται σε αυτή τη λέξη implosion. 5η Δεκεμβρίου η προθεσμία των τροπολογιών. Περιμένω τροπολογίες πολλές και καλές από πλευράς μας, ε, ακόμα και με λόγια πιο σκληρά από τα δικά μου. Και μετά θα έχουμε λίγο χρόνο, στον καινούριο πια χρόνο, να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Νομίζω ότι ε, η επόμενη συνάντηση θα είναι 23 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ κύριε Λόκεγκαρτ. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επανέλθει λίγο σχετικά με τις ερωτήσεις τις οποίες σας απίφθηνε ο κύριος Λόκεγκαρτ. Γιατί ο συνάδελφός σας από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου δεν έχει έρθει ακόμα. Να ζητήσω συλλογικά υπόψη για τους εκπροσώπους που έχουν λίγο καθυστερήσει, λέει η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκή Επιτροπής. Κοιτάξτε, εγώ δεν προβλέπω την αποκάλυψη για το Solvit. Αλλά πριν κάνουμε τις νέες συστάσεις, τα θέματα του Solvit τα συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη για την πιθανότητα υπογραφής ή δημιουργίας ενός κανονισμού. Εμείς θέλουμε ένα Solvit με συγκεκριμένες προθεσμίες. Θέλουμε ένα Solvit το οποίο να δουλεύει ε, γρήγορα. Αν βάλουμε ε, αν θέλετε το θέμα ας πούμε των 10 εβδομάδων μέσα σε ένα επίσημο νομικό δεσμευτικό κείμενο ε, πρώτα θα προσπαθήσω να βρω νομικά αν καλύπτομαι στα πλαίσια της προσπάθειας την οποία θα κάνω εγώ σαν εκπρόσωπος του Solvit για να λύσω ένα θέμα να μην κατηγορηθώ σαν σόλβιτ ότι δεν εφαρμόζω σωστά τον κοινοτικό νόμο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια κάποια στέρηση χρονική και δεν μπορεί να ληφθούν άμεσα υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία νομικά δεσμευτική όπως η διαδικασία της προσφυγής επί παραλήψη η οποία μπορεί να κρατήσει και χρόνια πολλά. Συνεπώς λοιπόν Εμείς δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα παρά μόνο αν μας ζητηθεί επίσημα να κάνουμε κάτι. Δεν είναι αυτή η λογική. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι δέκα εβδομάδες μπορεί να γίνουν μια, ένας χρόνος ή δέκα μήνες ε, και δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο αφαιρεί προς τη θέμενη αξία από το Σόλβιτ Και ακόμα και αν προσφύγει κανείς σε δικαστήριο, αυτό θα απαιτήσει πάρα πολύ ε, χρόνο. Η λέξη λοιπόν implosion και implode ίσως ήταν υπερβολική. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο ανεπίσημος χαρακτήρας των μεθόδων του Solvit επιτρέπει στα κέντρα Solvit να λύνουν τα προβλήματα γρήγορα, αποφεύγοντας την επίσημη ε, νομική κουζίνα. Επειδή έχω ασχοληθεί με το Solvit για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνω ότι εννοείται. Είναι δύσκολο, έχουν διαχειριστεί κάποιες υποθέσεις και ήταν αποτελεσματικά τα κέντρα Solvit, κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Ε, γεγονός είναι ότι υπάρχει μία απογοήτευση όταν το Solvit δεν μπορεί να λύσει κάτι, όπως λέει το όνομά του, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα νομικό εμπόδιο. Μπορεί να μην υπάρχει ε, το νομικό σύστημα από πίσω για να μπορέσει να λυθεί κάτι. Παρ' αυτά χρειαζόμαστε, όπως είπατε, να γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος ε, τι είναι το Solvit. Και ίσως είναι απλό αυτό. Πολλές ε, φορές το έχουμε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πει είχαν κληθεί τα μέλη της Επιτροπής μας ε, να ε, μπουν στο σύστημα ε, ως καταγγέλλοντες στο Solvit για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Νομίζω ότι αν τα, οι ευρωβουλευτές χρησιμοποιούν το Solvit για να λύσουν τα προβλήματά τους, τότε μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη θετική εμπειρία και στους υπολείπους. Πολύ σημαντικό αυτό. Να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο εισηγητής, ότι είναι πολύ ε, δύσκολο το χρονοδιάγραμμα. 5 Δεκεμβρίου, ως τις 5 Δεκεμβρίου για ε, τις τροπολογίες. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 9 Δεκεμβρίου, τις συμβιβαστικές στις 22 και θα ψηφίσουμε στις 23. Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε στην Ολομέλεια σύντομα, γιατί υπάρχει ολόκληρος κύκλος προετοιμασίας ε, για αυτό. Και ξέρετε ότι η τελευταία μας Ολομέλεια είναι τον Απρίλιο, οπότε, το, οπότε αν τον Ιανουάριο έχουμε ακόμη δουλειά, μας μένει μόνο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος. Πρέπει να έχουμε και μια σωστή συζήτηση για το θέμα αυτό, αν χρειαστεί. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει πίεση χρόνου και πρέπει να προγραμματίσουμε γέρος. Και σας το λέω αυτό για τις πολιτικές σας ομάδες. Πρέπει να τους περάσετε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα για όλους ε, όσους ε, παρακολουθούν στο ίντερνετ ε, ή δεν ήταν εδώ νωρίτερα. Αλλάξαμε την σειρά της ημερήσιας διάταξης. Τώρα θα ασχοληθούμε με την έκθεση Αρίας Ετσεβερία για την ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και, και μεγάλη προτεραιότητα. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νέα χρονοδιαγράμματα ή θα έχει νέα χρονοδιαγράμματα σύντομα. Οπότε να ζητήσω από τον Παύλο Αρίας να μας μιλήσει για τις συμβιβαστικές τροπολογίες είναι εδώ η κυρία Σενάλοβα, καλώ ήρθατε και πάλι. Ο κύριο Κρόιτσμαν είναι εδώ, ο Ρούλε. Ο κύριος Μπίλαν δεν είναι εδώ. Α, μόλι ήρθε ο κύριος Μπίλαν. Οπότε υπάρχει ε, μια πλήρη ομάδα σκιωδών εισηγητών. Πρώτα ο κύριος Άρια. Άριας. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία για το διάλογο που είχαμε αυτούς τους μήνες με τους χειώδεις εισηγητές στη διαδικασία εκπόνησης αυτής της έκθεσης καθώς επίσης και με τις τροπολογίες, για τις τροπολογίες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο αυτού του χαρτοφυλακίου και τη γενική συνένεση στην οποία καταλήξαμε οι κυριότερες ομάδες για τα πιο σημαντικά στοιχεία. Επίσης θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να παραστώ στην ανταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες των προηγούμενο μήνα. Μία νέα, ας το πω έτσι, ε, θεραπεία ε, με ανάγκασε να απουσιάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον συνάδελφο που έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει εκπροσώπηση εξ ονόματός μου και τον κύριο Σβάμπ που με ξεπροσώπησε τότε. Όπως τότε εξ ονόματός μου μίλησε και είπε ο συνάδελφος Σβάμπ τότε, οι περισσότερες τροπολογίες θεωρώ ότι είναι θετικές και συνεισφέρουν να εμπλουτίσουν και να συμπληρώσουν την έκθεση. Γι' αυτό θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Επίσης όλους τους ευρωβουλευτές που κατέθεσαν τροπολογίες που εμπλουτίζουν το κείμενο όπως ιδιαίτερα τον κύριο Κορέεντε Κάμπος και την κυρία Γκέπαρντ. Για την πλειοψηφία αυτών των τροπολογιών ζητώ θετική ψήφιση αυτών των τροπολογιών. Για άλλα, ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση και συζήτηση επ' αυτών και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στις αναγκαίες συμφωνίες ώστε αυτή η τόσο σημαντική έκθεση να μπορέσει να ευδοκιμήσει, να εγκριθεί. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το πιο σημαντικό θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί έναν κύριο πυλώνα για την ολοκλήρωση ε, της εσωτερικής αγοράς. Ολόκληρη την κοινοβουλευτική θητεία εργαζόμαστε επ' αυτού του στόχου. Οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις όπως και άλλες επιχειρήσεις χρειάζονται έναν ολοκληρωμένο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, παράδοση θεμάτων. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξη ε, και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και όπω είδαμε στι προηγούμενε συναντήσει με του σκιώδει συζητητέ, μπορώ να πω ότι οι διάφορε πολιτικέ ομάδε συμφωνούμε στα διάφορα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προαγάγουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό εφικτό, δουλέψαμε πολύ σε αυτή την Επιτροπή, όπω όλοι γνωρίζουν. Ήδη το εγκρίναμε την έκθεση ολοκληρώνοντας ε, τις προτάσεις για την ενιαία εσωτερική αγορά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συμπληρώνοντας και με το ψηφιακό εμπόριο και από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα είχαμε συνολικά 16 συνεδριάσεις ομάδων εργασίας για ε, ψηφιακή, το ψηφιακό εμπόριο και την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ευρώπη. Και εγκρίναμε αυτές τις δυνατότητες τον προηγούμενο Ιούλιο και τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών και η εναλλακτική επίλυση ε, διαφορών και τριβών online ηλεκτρονικά ψηφιακά ήταν ένα σημαντικό βήμα. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι ένα από τα κλειδιά της ψηφιακής αγοράς. Θα έλεγα ότι είναι είναι θεμελιώδες κλειδί αυτή της αγοράς. Πρέπει να προαχθεί για να δώσουμε αυτή την προώθηση και να διατηρήσουμε αυτή την προώθηση ώστε να υπάρξουν τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Υπό αυτή την προσέγγιση ε, συνέταξα διάφορες τροπολογίες και πρότεινα συνολικά οκτώ συμβιβαστικές τροπολογίες σε διαφορετικούς τομείς που είναι σημαντικοί όπως ε, η αύξηση για παράδειγμα των δυνατοτήτων σε σχέση με τους καταναλωτές, η ενημέρωση, βελτίωση, η βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων να μελετήσουμε την βιωσιμότητα ώστε να υπάρξει ακριβώς ε, ένα σύμβολο, ένα έμβλημα αξιοπιστίας ε, για την Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα. Να αυξήσουμε και την ελαστικότητα των υπηρεσιών αποστολής διασφαλίζοντας τους όρους απασχόλησης που καθορίζονται από την ομοθεσία κρατών μελών. Για άλλες τροπολογίες που δεν, άλλα θέματα που δεν εντάσσονται σε αυτούς τους συμβιβασμούς <clears throat> και που θεωρώ ότι και αυτές είναι θετικές τροπολογίες θα ζητήσω να υπερψηφιστούν αλλά δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε αυτούς τους συμβιβασμούς όπως είναι οι τροπολογίες του κυρίου Χορέια Ντεκάμπος 2, 3, 5, 7, 12, 25, 26 του κυρίου Μπίλαν οι 45 και 48 του κυρίου Κρότσμαν οι 17, και 59 της ε, κυρίας Σιναλόβα, Εύελιν Γκέπατ και επιπλέον πάλι του κυρίου Κορέιντε Κάμπος για την ενδυνάμωση, την ένταση ή την δημιουργία webs, δικτύων για σύγκριση τιμών για αυτές τις υπηρεσίες αποστολών οι 19, 20 και 47 τροπολογίες. Αυτά σε γενικές γραμμές είχα να πω είναι οι κυριότερες γραμμές που ήθελα να σχολιάσω τώρα. Ολοκλήρωσα. Είμαι στη διάθεση να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις των συναδέλφων και να ανταλλάξουμε απόψεις. απόψεις. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τις συμφωνίες που είναι αναγκαίες για την έγκριση της έκθεσης με την υποστήριξη όλων των ομάδων. Ευχαριστώ για το έργο που επιτελέστηκε από αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτή η κοινοβουλευτική θητεία οδήγησε στο να αφυπνιστεί η ψηφιακή Ευρώπη πιστεύω. Και είμαι βέβαιο αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία δίνοντας περαιτέρω βήματα, κάνοντας περαιτέρω βήματα προ ε, προς το μέλλον για να βελτιωθεί η κατάσταση και να υπάρξει πρόοδο. Ευχαριστώ. Good. thank you very much indeed. Ευχαριστώ. Πράγματι έρχεται σε σωστή στιγμή η πρόταση αυτή. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία και από την ομάδα εργασία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη που δεν καλωσόρισα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πριν. Θα σας δώσω το λόγο ε, ε, λίγο αργότερα. Ας ακούσουμε όμως πρώτα τους σκιώδους της ηγητές. Η κυρία Σανάλοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον κύριο Τσεβερία για τις συμβιβαστικές προτάσεις. Παράλληλα να πω ότι δυστυχώς εγώ πήρα το κείμενο αυτό χθε το απόγευμα και δεν είχα χρόνο για να το συζητήσω και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έκανα όμως μια, μια βιαστική, αν θέλετε, εξέταση των συμβιβαστικών προτάσεων και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένα σχόλια εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας των σοσιαλιστών. Ε, δεν μπορούμε εμείς να αποδεχθούμε οι τροπολογίες ε, οι οποίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας ε, στα πλαίσια της παράδοσης δεμάτων να μην είναι τόσο πλήρης όσο θα θέλαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα της συζήτησης και η συμβιβαστική πρόταση αφορά μόνο το προήμιο. Η συμβιβαστική πρόταση 1 λοιπόν δεν αντικατοπτρίζει δυστυχώς τις προτεραιότητές μας. Ως έχει λοιπόν θα προτείναμε εμείς να ε, υπάρξουν αλλαγές. Ο εισηγητής αναφέρθηκε και σε κάποια επιμέρους θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα στις συμβιβαστικές προτάσεις. Στα πλαίσια της 1 σαν παράδειγμα τι γίνεται με τις τροπολογίες 32, 33 και 35, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τροπολογία 1. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι κάτι το οποίο έχω επανειλημμένα θέση. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ετικέτας εμπιστοσύνης. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει ε, πάρα πολύ πιθανότητα προστιθέμενης αξίας, ε, εγγύηση ποιότητας, διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους εισηγητές για τη συμβιβαστική πρόταση υπαριθμών 7. Και εδώ βέβαια θα μπορούσε να είναι ο κύριος Ετσεβερία πιο φιλόδοξος λίγο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες της στον τομέα της ετικέτας εμπιστοσύνης. Θα προετοιμάσουμε περαιτέρω λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις και θα τις διανύμουμε γραπτά σε όλους τους συναδέλφους για να τις λάβουν υπόψη. Ελπίζω, πιστεύω μάλλον ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε από πλευράς της πολιτικής μας ομάδας την πρόταση Ετσεβερία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος Κρόιτσμαρκ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, θετικότατες ε, συμβαστικές τροπολογίες στον εισηγητή. Υπό τη σημερινή μορφή όλες αυτές τις προτάσεις μπορώ να τις υποστηρίξω και για τις ε, δραστηριότητες ε, των επιχειρήσεων ε, που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την νομοθεσία και να την σέβονται όπως και σε άλλους τομείς. Η δυναμική ανάπτυξη της αγοράς παράδοσης δεμάτων πρέπει να έχει και την κοινωνική διάσταση. Όμως οι διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές και πολιτιστικές παραδόσεις πρέπει να είναι σεβαστές. Δεν πρέπει όλα να επαναρρυθμίζονται. Γι' αυτό ευχαριστώ τον εισηγητή που λαμβάνει υπόψη αυτή την πτυχή και τον την πρότασή μου στο συμβασμό 5 την ενέταξε συμβαστική τροπολογία. Οι επιχειρήσεις πρέπει με βελτιστοποιημένες διαδικασίες να μπορούν ε, να απλουστεύσουν ε, την παράδοση πολλών ε, μικρών αποστολών. Όπως και στην τελευταία συζήτηση τόνισα, υποστηρίζω καταρχήν την πρόταση του εισηγητή να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σήμα ως μάρκα, ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας, παρότι αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την παράδοση πακέτων, παράδοση δεμάτων. Χαιρετίζω επίσης την πρόταση υπαριθμών 7 ως συμβιβασμό διότι <clears throat> σε σχέση με τα κριτήρια δεν, δεν πρέπει να επιβαρύνεται η διαδικασία αυτής της μάρκας, αυτού του συμβόλου ε, με υπερβολικές ρυθμίσεις. Πρέπει η ποιότητα να διασφαλίζεται. Η τήρηση αυτών των διατάξεων πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο. Επιπρόσθετα οικολογικά, κοινωνικά κριτήρια νομίζω θα ήταν υπερβολικά η τήρηση όλων των κριτηρίων πρέπει και κρατικά να επιτηρείται Όσο πιο περίπλοκες είναι οι απαιτήσει, τόσο πιο δαπανηρή η έλεγχη. <clears throat> Γι' αυτό σε σχέση με τους ε, συναδέλφους ε, θα ήθελα να ζητήσω να αποφύγουμε την γραφειοκρατική επιβάρυνση. Σημερίζομαι την εκτίμηση στο Συμβασμό 8 ότι όλα τα νομοθετικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά ώστε να μην περιοριστεί η δυναμική ανάπτυξη του τομέα. Μόνο στην τελευταία πρόταση με την πρόταση του κυρίου Σβάπ θα ήθελα μια μικρή παρατήρηση να κάνω η επιτήρηση αγορών. Αποκινούμε τη διασφάλιση, διαπίστωση όταν υπάρχει κάποια αποτυχία της αγοράς. Όταν κάνουμε λόγο για επιτήρηση, τότε τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν τις νομικές ε, διατάξεις ε, και να μεριμνούμε γι' αυτό. Ίσως λοιπόν έτσι θα μπορούσε ο κύριος Σβάμπ αυτό να το ε, διευκρινίσει για να είναι πιο ε, αποτελεσματικό. Θα έπρεπε όμως ε, να έχουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρόιτσμαν. Κύριε Ρούλα. Λοιπόν, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να πω στον προλαλήσαντα, το βρίσκω αξιοπερίεργο αυτό το αίτημα, γιατί δεν καταθέσαμε εμεί τροπολογίε κύριε Κρότσμαν. Εντάξει, ίσως να το σημειώσετε αυτό, όπου η ενεργειακή επίδοση σε αυτόν τον τομέα, η ενεργειακή απόδοση διαδραματίζει ρόλο, αλλά δεν πρέπει αυτό ξεχωριστά να το εξετάσουμε. Πρέπει γενικά με την ε, ανάπτυξη, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ε, στην Ευρώπη να το εξετάσουμε. Καταρχήν οι ε, συμβαστικές τροπολογίες βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά με τις διατυπώσεις πρέπει και εγώ να πω ότι πρέπει να τις εξετάσω τις προτάσεις αυτές σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Μπίλαν, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω από πλευρά μου να σχολιάσω σύντομα τι συμβαστικέ τροπολογίε, τη συμβαστική τροπολογία 5 και την 8. Αφορούν και τροπολογίες που εγώ κατέθεσα. Μπορώ να υποστηρίξω αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Πολύ καλά αντανακλούν και τις δικές μου προθέσεις. Τώρα, για το συμβιβασμό 1 για την κοινωνική διάσταση σε αυτό το ζήτημα προτάθηκε πολλές φορές ε, στο παρελθόν ε, και από τους σοσιαλιστές με, τροπολογίε με τροπολογίες τους. Νομίζω καλά αντανακλώνται οι ιδέες αυτές ε, στη συμβαστική τροπολογία του εισηγητή παρότι, ότι, παρότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες θα έπρεπε στην Επιτροπή Ανάπτυξης να εξεταστούν και πιστεύω ότι θα μπορέσω τελικά να υπερψηφίσω αυτό το συμβιβασμό παρότι δεν καλύπτει απόλυτα 100%. Όμως για την αξιόπιστη ευρωπαϊκή αγορά για μια, ένα σύμβολο αξίζει νομίζω να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μάρκα, ένα σύμβολο που θα μπορούσε να εισαχθεί για την αξιοπιστία των υπηρεσιών Ενώσεως στην Ευρώπη. Αυτό τι θα, πώς θα λειτουργεί, θα δίνεται σε εθνικές ε, επιχειρήσεις και εταιρείες ή και εθνικές κρατικές εταιρείες θα μπορούσαν και αυτές σε κρατικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Θα υποστηρίξουμε αυτές τις τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε για αυτό το έγγραφο. Thank you. Now, does anyone else... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες. Θέλει κανείς άλλος ε, να πάρει το λόγο. Μόλις πρόσεξα για τη συμβιβαστική τροπολογία ε, να πρέπει να δείτε λίγο τη διατύπωση, γιατί λέει εδώ στα αγγλικά ότι η κατάλληλη εκπαίδευση είναι σημαντική για την επίτευξη ε, της ανεργίας. Μου φαίνεται ότι Κάτι άλλο θέλατε να πείτε. Δεν νομίζω να θέλετε να πείτε κάτι τέτοιο. Κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ στη διατύπωση. Θέλετε να, ε, να επιτύχετε υψηλού επίπεδου ε, απασχόληση και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Μάλλον αυτό θέλετε να πείτε. Κυρία Λαμότ, μήπως θέλετε να πάρετε το λόγο. Είδα και τη συνάδελφό σας εχθές ε, που μου είπε ότι επεξεργάζεστε έναν χάρτη πορείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που ο κύριος Βερνέρ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Είναι σε αποστολή. Λείπει. Εδώ και κάποια χρόνια στην ε, ενιαία ψηφιακή αγορά και ειδικότερα ως προς το θέμα αυτό των, ε, των, ε, της παράδοσης πακέτων καταρχάς να ευχαριστήσω τον Άρια Σετσεβερία, τον εισηγητή για τη δουλειά του. Υπήρξε μια σύγκληση απόψεων λοιπόν από την αρχή των εργασιών αυτών και διαπίστωσα ότι Πιο συγκεκριμένα αναφερθήκατε στα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στο επίκεντρο των εργασιών μας, τα κοινωνικά ε, ζητήματα, ε, τα οποία βεβαίως είναι πολύ ευαίσθητα στον τομέα αυτό. Είναι σαφές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εξέλιξη του τομέα παράδοσης ε, δεμάτων πρέπει να γίνει βέβαια στο πλαίσιο του, του διαλόγου του κοινωνικού, πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων προχωρούμε κι εμεί ε, παράλληλα με τις δικές σας εργασίες. εργασίες ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το χάρτη πορεία που αναφέρατε πριν από τις ε, διακοπέ των Χριστουγέννων. Ένας χάρτης που θα συμπεριλάβει, υποθέτω, το σύνολο των ε, ετοιμάτων σας. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειε βεβαίως σήμερα δεν ε, θα επιβαρύνει περαιτέρω και τη γραφειοκρατία γιατί έχουμε προτείνει μια μη ρυθμιστική διαδικασία η οποία συνοδεύει τις επιχειρήσεις ε, με μια παρακολούθηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να μας ικανοποιεί νομίζω εδώ και κάτι παραπάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου. Το επεξεργαζόμαστε, το δουλεύουμε. Ξεκινήσαμε από μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε ιδιαίτερη συνένεση όταν μιλούσαμε με τον κλάδο. Υπήρχαν ε, όμως προβλήματα. Και τώρα έχει δημιουργηθεί μια όθηση για να το πω όπως το είπε και ο εισηγητής. Ε, αρχίζουν σιγά σιγά οι εταίροι να μετακινούνται ε, ως προς τις απόψεις τους και νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την όθηση και να την πλαισιώσουμε, για να το πω έτσι. Ελπίζω λοιπόν πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές να υπάρξει ο χάρτης πορείας που σας δείξει ακριβώς ε, ποιες είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με άξονες ε, την πληροφόρηση των καταναλωτών, τη βελτίωση της ποιότητας, ε, την τιμολόγηση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και στη συνέχεια προσπάθειες επίλυσης υπέρ του καταναλωτή όταν υπάρχουν προβλήματα και δεν πάνε καλά τα πράγματα σε σχέση με την παράδοση ενός δέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με χαρά βλέπω ότι το θέμα παρακολουθείται σωστά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε ιδέες που να καταστήσουν τη διαδικασία αυτή της παράδοσης πιο αποτελεσματική, πιο αξιόπιστη σεβόμενοι τον ανταγωνισμό αλλά καθιστώντας εύκολη και την πρόσβαση στον τομέα για τις μικρές εταιρείες οι οποίες παρέχουν τον απαιτούμενο δυναμισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια συνάντηση που ήμουν χθε, μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις είπαν ότι προσφέρουν κάποιες απλές μορφές παράδοσης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χωρίς ε, ίσως την δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας επίδοσης, παράδοσης μάλλον. Ε, κι όμως και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους μέσα τεχνολογικά. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή, θέλετε, ε, ε, κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι ή Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σημείωσα πολύ προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν και θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από αυτές τις παρατηρήσεις. Η πρόθεση του εγγράφου χωρίς αμφιβολία είναι να βελτιώσει τις υπηρεσίες αποστολής μέσω ελαστικοποίησης και απλούστευσης. Λοιπόν, εγώ σε σχέση με την παρέμβαση που έκανε η κυρία Ρανόβα, πρώτον θέλω να την ευχαριστήσω για το έργο που αφοσίωσε, αφιέρωσε σε αυτό το θέμα. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι συμφωνούμε όσον αφορά το έργο που επιτελέσαμε και τους στόχους μας. Πολύ περισσότερο συμφωνούμε από ό,τι θεωρεί εκείνη. Εγώ ειλικρινά δεν είμαι καθόλου κατά των τροπολογιών που ετέθησαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εκείνο όμω το οποίο δεν μπορώ να δω είναι πως ένα έγγραφο που έχει 17 παραγράφους μπορεί 30 παραγράφους να συμπεριλάβει για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει μια ξεχωριστή κοινοβουλευτική επιτροπή για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η Επιτροπή Επασχόλησης. Έτσι λοιπόν πιστεύω δεν έχει νόημα να εντάξουμε 30 παραγράφους, 30 εδάφια για αυτό το θέμα στην έκθεσή μου. Και εγώ πρέπει να πω και το λέω με κάθε διαφάνεια και ειλικρίνεια, κάπως είμαι κατά της ε, ένταξης ε, αυτών των προτάσεων σε μια συμβαστική τροπολογία. Δεν ήταν η θέση σε μια συμβαστική τροπολογία γι' αυτό. Μετά όμως ε, το ξανασκέφτηκα αυτό, συζήτησα με συναδέλφους και καταλήξαμε ότι σε μια τροπολογία συμβιβαστική μια και δεν θα μπορούσα να είμαι εναντίον, θα μπορούσε ίσως να γίνει αυτό. Και έτσι λοιπόν στο συμβιβασμό ένα μπορούσε να, συμβιβα... να ενταχθεί αυτό. Αν νομίζει η σοσιαλιστική ομάδα ότι αυτό δεν επαρκεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν αληθεύει. Πολύ σωστά νομίζω μπορεί έτσι να διαφοροποιηθούν τα πράγματα σε σχέση με τις προτάσεις ε, που έχουν υποβληθεί. Και έτσι αν θέλετε αυτό να συμπεριληφθεί στην έκθεση, νομίζω ότι είναι το ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε και θα ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους, ώστε όλοι μας να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο συμβασμό όπως αυτόν. Υπάρχουν επίσης και κάποιες, κάποιοι δισταγμοί όπως ακούσαμε για αυτή την, ε, για αυτή την ε, διαμόρφωση αυτής της συμβαστικής τροπολογίας 1. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ίσως αληθεύει ότι δεν είναι επαρκή η 7 δεν είναι ίσως ε, η πιο ευρεία ε, φιλόδοξη τροπολογία, συμβιβαστική τροπολογία. Όμως σε όλο το έργο που κάναμε για το σύμβολο ποιότητας έχει συμπεριληφθεί στις εκθέσεις και εδώ και χρόνια εργαζόμαστε ως εισηγητές και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει αυτό το, να επιτελέσει αυτό το έργο, να επιτευχθεί αυτό το σύμβολο, αυτή η μάρκα ποιότητας και αξιοπιστίας. Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο ε, μπορεί να προχωρήσει και έτσι λοιπόν η συμβαστική αυτή τροπολογία εκφράζει με κάθε σαφήνεια ποιοι είναι οι στόχοι μας για αυτό το trust το, τη μάρκα ποιότητας, τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το πετύχουμε. Για τον κύριο Κρόισμαν που και αυτόν τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του και φυσικά επίσης και για όλα όσα πρότεινε και συνεισέφερε. Πιστεύω ότι και για τους σκιώδεις εισηγητές προσπάθησαν και αυτό είναι ο στόχος ο τελικός, να εμπλουτίσουν το κείμενο έτσι και να το βελτιώσουν. Και υπό αυτή την πρόπτικη έλαβα υπόψη τις τροπολογίες αυτές όσες μπορούσαν να ενταχθούν σε συμβαστικές τροπολογίες. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόμαστε για να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο έργο και στους στόχους μας. Είναι η ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων και της οικονομίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να βελτιωθούν οι παραδόσεις δεμάτων και όσον αφορά τις, πι... τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και για τους καταναλωτές γενικότερα και τις επιχειρήσεις. Ο συμβιβασμό 5 κάνει λόγο ακριβώς γι' αυτό. Για το θέμα του συμβιβασμού 7. Επανερχόμαστε στην τροπολογία τη συμβιβαστική για το θέμα του, της μάρκας ποιότητας, του συμβόλου ποιότητας, τρασμάρκα. Είναι κάτι που θα μπορέσουμε να ξαναδούμε στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε σε δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, στο Στρασβούργο. Όπου έτσι δεν είναι η επόμενη ε, συνάντηση των ε, ε, παϊόντων και έτσι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά αυτή την προσπάθεια. Το αντίθετο, πρέπει να υπάρξει ελαστικοποίηση, απλούστευση στο μέτρο του εφικτού. Και για το συμβιβασμό 8, η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ πολύ με αυτά τα οποία αναφέρονται. Για τις τροπολογίες 4 και 5 θα συζητήσουμε με τον κύριο Σβάμπ να δούμε αν έγινε κατανοητό απόλυτα αυτό το οποίο στοχεύει να ε, πει ο κύριος Σβάμπ με αυτές τις τροπολογίες Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Σβάμπα θα, είναι απόλυτα, θα έχει ανοιχτό πνεύμα να συζητηθούν αυτά τα θέματα μαζί σας ή να δοθούν όποιες επεξηγήσεις χρειάζονται. Για το θέμα το χρονικό, εμείς όπως και σε όλο το έργο της Επιτροπής, ο χρόνος δεν περισσεύει, πιέζει ο χρόνος και για τις συμβαστικές τροπολογίες ε, ε, όταν ήταν δυνατόν ε, για την, να συνταχθούν και να αποσταλούν. Δεν είναι το, η μόνη έκθεση που αντιμετωπίζει πρόβλημα χρόνου. Ζητώ συγγνώμη για τα προβλήματα για να υπάρξει δυνατότητα να, να εξεταστούν και να συζητηθούν και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και ζητώ συγγνώμη για τα προβλήματα. Για τον κύριο Μπίλαν ευχαριστώ για τα σχόλιά του. Για την τροπολογία 1 επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι είναι μια καλή τροπολογία λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της σοσιαλιστικής ομάδας. Και λοιπόν <clears throat> αν θα ήταν υπέρ της διατήρησης αυτού του συμβιβασμού και να υποστηρίξουν αυτό το συμβιβασμό νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και πολύ θετικό για όλους. Τώρα, για το σύμβολο ποιότητας, το έμβλημα ποιότητας, για τον συμβιβασμό 7 εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ε, μια μάρκα για όλους, ένα σύμβολο για όλους που θα ίσχυε για όλα και για όλους. Όμως καθορίζουμε κάποιες γενικές γραμμές για να προσπαθήσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την... Ε, και τα θεσμικά όργανα να ε, μπορέσουν να δράσουν ώστε να μην χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση εδώ Υπάρχουν ανοιχτά εγχειρήματα και κλειστά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή, να υπάρχει πρόσβαση για όλους σε, αυτό το, σε αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα του Προέδρου Χάρμπορ. Θα δούμε αν είναι θέμα μετάφρασης ή όχι ή αν είναι θέμα διατύπωσης. Ευχαριστούμε για αυτή την επισήμαση και θα δούμε το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η ψήφιση, αν θυμάμαι καλά, 17 Δεκεμβρίου θα γίνει, έτσι, στην Επιτροπή μας. Στην, ε, ομάδα μας. Και θα έχουμε και μια συνάντηση όπου θα είχα να, ήθελα να ζητήσω να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Και με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ε, γνωρίζετε σε σχέση με αυτή τη συνεδρίαση. Ελπίζω ότι εκεί θα μπορέσουμε να συνέλθουμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τις συμβαστικές τροπολογίες και όλα τα ανοιχτά θέματα. Ευχαριστώ. yes, well, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Πράγματι το χρονοδιάγραμμα λέει ψηφοφορία στις 17 Δεκεμβρίου. Εδώ παρατηρώ ότι οι αρμόδιες επιτροπές ε, και μεταφορών και απασχόλησης θα αποφασίσουν στις 6 Δεκεμβρίου, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να τα εξετάσετε αυτά ε, στο Στρασβούργο. Μπορείτε να λάβετε υπόψη τις θέσεις τους ε, και τις επιτροπές υπεύθυνες για θέματα αγνομοδότησης και η κυρία Σενάλοβα είναι δραστήρια στην Επιτροπή Μεταφορών και θα μας βοηθήσει ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ε, πράγματι είναι σε εύθετο χρόνο έρχεται η συζήτηση της έκθεσης αυτής. Νομίζω θα υπάρξει και μια κάποια δημοσιότητα γιατί ε, το πράσινο ε, βιβλίο σε εισαγωγικά σε σχέση με την παράδοση δεμάτων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της φροντίδας μας για τους καταναλωτές. Περνάμε σε ένα άλλο τώρα σημαντικό θέμα, σημαντικό για τους πολίτες. Είναι ένας τομέας ο οποίος θα πρέπει να μας αφορά. Πρόκειται για το θέμα της προσβασιμότητας στους ιστοτόπους του δημοσίου. Αλλάξαμε τη σειρά της συζήτησης αυτό κανονικά θα έπρεπε να το συζητήσουμε νωρίτερα, αλλά χαίρομαι που έχουμε τον κύριο Χατζημαρκάκη μαζί μας. Έχουμε λοιπόν μισή ώρα για να συζητήσουμε τα των συμβιβαστικών τροπολογιών. Η Επιτροπή αργεί λιγάκι σήμερα, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε εφόσον το θέλει ο εισηγητής και θα επανέλθουμε στο θέμα. Υπάρχουν 30 συμβιβαστικές ο ε, κύριος Τρασκόφσκι, ένας από τους εισηγητές για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έγινε υπουργός, υπουργοποιήθηκε στην Πολωνία, θα πρέπει να τον συγχαρούμε για την απουσία του. Αυτό είναι πολύ καλό νέο για την Επιτροπή μας και θα αναλάβει τη θέση του ο κύριος Φάμπα. Ο κύριος Μπίλαντ είναι εδώ, ο κύριος Ένστρομ είναι εδώ, θα υπάρξει αντικατάσταση ε, αν κάποιος είναι απόν, οπότε μπορείτε να παρουσιάσετε τις συμβιβαστικές σας κύριε Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ. Πράγματι ο κύριος Χατζημαρκάκης ήταν ένα από τα πιο, ε, αν θέλετε, σημαντικά μέλη στην διαδικασία αυτή. Κρίμα που θα φύγει, αλλά θα μείνει μαζί μας μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και μετά μπορεί να συνεχίσει να πιέζει γύρω από το θέμα αυτό σαν υπουργό γιατί θα είναι υπεύθυνο για την ψηφιακή ατζέντα. Είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στις αρμοδιότητές του και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θα επανέλθω στα της διαδικασίας. Η οδηγία αυτή όπως ξέρετε έχει σαν στόχο να καταστήσει όλες τις ιστοσελίδες του δημοσίου προσβάσιμες για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι δεδομένες αυτές οι υπηρεσίες, αλλά έχει σημασία να μην αποκλείεται κανείς από τη διαδικασία αυτή και δεν αναφέρουμε μόνο στους αναπήρους αλλά και στους ιδιαίτερα ηλικιωμένους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, ακούσαμε την άποψη πολλών πλευρών και της βιομηχανίας και των καταναλωτών και της ομάδας η οποία φύγεται, αν θέλετε πιθανώς από τη διαδικασία αυτή, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας που παρακολουθούν από κοντά αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους ορισμούς. Έχουμε ε, μείνει, αν θέλετε, πάρα πολύ κοντά στα παγκόμια standards και έχουμε ευθυγραμμίσει κατά κάποιο τρόπο τις διαδικασίες που οδηγούν στην διατύπωση των ορισμών έτσι ώστε να είμαστε ε, απολύτως συμβατοί με τις διεθνώς ισχύουσες ρυθμίσεις. Δεύτερο βασικό θέμα είναι η εμβέλεια αυτής της ε, προτινόμενης ρύθμισης. Και αυτό συζητήθηκε εξ αρχής, το πιο, ε, είναι το πιο κρίσιμο θέμα. Ποια είναι η εμβέλεια, τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, και εμείς εδώ αποκλίναμε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στο νέο περιεχόμενο ή το τροποποιημένο νέο περιεχόμενο και το παλαιό περιεχόμενο. Δεν ακολουθήσαμε την γραμμή η οποία λέγει ότι υπάρχει απλά ένας κατάλογος θεμάτων και υπηρεσιών τις οποίες θα πρέπει να παρέχουν τα κράτη-μέλη. Όχι, κάθε νέο περιεχόμενο ψηφιακό από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ψηφιακά. Το παλαιό περιεχόμενο πρέπει να γίνει διαθέσιμο ψηφιακά από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Ακούγεται φιλόδοξο, είναι φιλόδοξο, είναι όμως και εφικτό. Πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο για τη σωστή εφαρμογή αυτής της πρότασης. Σχετικά τώρα με το ποιόν του περιεχομένου υπάρχει μια παραδοσιακή μεταβατική περίοδος. Τώρα, τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται όχι από το, όχι από το κράτος, από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές, ε, ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει ε, μία προσθήκη η οποία ε, εξηγεί ακριβώς ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες παρεχόμενες μεν από τις ιδιωτικές υπηρεσίες πρέπει, ε, οφείλεται όμως να παρέχονται ψηφιακά. Εμείς κάνουμε τρεις βασικές λειτουργίες αν θέλετε, την παρακολούθηση, ε, καταρχάς σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ορίσουν μια αρμοδία επί του θέματος αρχή επί τη βάση της εφαρμογής της αρχής επικουρικότητας. Δεύτερον είναι ο μηχανισμός παραπώνων και να αναφέρονται τα κράτη-μέλη σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού. Και τρίτον είναι ε, η εφαρμογή πλήρω του συστήματος, η παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος. Σε όλες τις πολιτικές ομάδες έχει υπάρξει μια κάποια συνένεση θα έλεγα ε, με τη διαδικασία αυτή. Έχουμε 30 συμβιβαστικές τροπολογίες. Πρόεδρε, πράγματι δουλέψαμε σκληρά και τα μέλη αλλά και η γραμματεία, η κυρία Μπρίγκετ Χάρτ που είναι εκεί μαζί σας, έκανε τεράστιες προσπάθειες. Συνολικά έχουμε 240 τροπολογίες, αλλά οι 30 συμβιβαστικές νομίζω καλύπτουν ε, σχεδόν όλες τις τροπολογίες των συναδέλφων. Λάβαμε υπόψη τα σχόλια από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι για αύριο περιμένουμε ένα σωστό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Θα έχουμε μια ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να βασίσουμε την διαπραγμάτευση. Αυτό έχει σημασία ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα έλεγα είναι ένα εύκολος, ένα εύκολο φρούτο ε, για, τα, για την επόμενη Προεδρία. Υπάρχουν δύσκολα θέματα γύρω από το ψηφιακό τομέα όπως οι παρακολουθήσεις, οι μυστικές κτλ. Και ενώ αυτό αντίθετα παρέχεται με πολύ μεγάλη ευκολία στην πολιτική εξουσία και γι' αυτό θα ήθελα να σας παροτρύνω να περάσουμε σε συμφωνία στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης. Αύριο μετά την ψηφοφορία να συζητήσουμε το θέμα με την ομάδα εργασίας της Λιθουανικής Προεδρίας, να το συζητήσουν και αυτοί πρώτα βέβαια, έτσι ώστε όλες, όλοι οι μηχανισμοί που έχουμε ε, στη διάθεσή μας ε, και σε σχέση με την Προεδρία και σε σχέση με τον μεγάλο αδελφό την Γερμανία στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχουν εξαντληθεί έτσι ώστε οι Έλληνες που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου να μας οδηγήσουν ε, στο κλείσιμο του θέματος με ένα στόχο. Τον Φεβρουάριο σε μία από τις δύο Ολομέλειες να ψηφίσουμε σαν Κοινοβούλιο. Και αυτή είναι και η τελευταία δυνατότητα γιατί αν ψηφίσουμε μετά από το Φεβρουάριο τότε πλέον αυτό το φρούτο ναι μεν βρίσκεται χαμηλά αλλά κανείς δεν μπορεί να το κόψει. Έχουμε λοιπόν εμείς συζητήσει επί τη βάση των συμβιβαστικών προτάσεων έχει υπάρξει μια, ένα θετικό πνεύμα, είναι θετικό το πνεύμα και από πλευρά της Προεδρίας και ο κ. Στρασκόφσκι, ο νέος υπουργός επ' αυτών των θεμάτων στην Πολωνία, ε, ε, θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ επίσης ε, και τον κύριο Γκασιαραμών, όπως επίσης και τον κύριο Έγκστρομ, που έχουν και αυτοί βοηθήσει πολύ στις τελικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ επίσης και για την παρουσίαση των συζητήσεων που είχατε με την Προεδρία που παίζει σημαντικό ρόλο βέβαια. Βρισκόμαστε σε μια καλή φάση πλέον έτσι ώστε να υπάρξει ψηφοφορία όπως και όταν πρέπει. Και να υπάρξει και πιο πριν μια κατάλληλη εντολή διαπραγμάτευσης. Ας ακούσουμε τώρα τις απόψεις των, των σκιωδών. Ο κύριος Σφάμπ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν, τους συναδέλφους των φιλελευθέρων και τον κύριο Χατζημαρκάκη ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία. Πολλά από αυτά που πρότεινε απόλυτα βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση και πρότειναν. Θέλω <clears throat> και να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Τσασκόφσκης και όδηση που όπως είπατε σωστά <clears throat> διορίστηκε ως υπουργό στη νέα <clears throat> πολωνική κυβέρνηση για ψηφιακά θέματα ακριβώς. Και έτσι σίγουρα θα, είναι, θα μας συνοδεύσει και μας υποστηρίζει σε αυτό το θέμα. Μετά όμως ε, από το Δεκέμβριο θα, ε, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα από πλευράς του. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε όλα τα όσα μας ανέφερε ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, από πλευράς μας. Τι συμβαίνει εδώ. Τα, τις τελευταίες εβδομάδες κάποια πολύ επίμαχα θέματα για συμβαστικές τροπολογίες μπόρεσαν να επιληθούν. Και έτσι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις τριβές και διαφορές μεταξύ μας. Υποστηρίζουμε το στόχο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο προσβασιμότητα ή στο προσπελασιμότητα <clears throat> όσον αφορά κράτη κρατικές υπηρεσίες ε, και θεσμούς να είναι με τέτοιο τρόπο η διαμόρφωση αυτών ώστε να υπάρχει πρόσβαση για όλους τους χρήστες και να διασφαλίζουμε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι πληροφορίες να μπορούν να καταλήγουν στους πολίτες και να χρησιμοποιούνται από αυτούς. Κυρίως πρέπει να προσέξουμε οι πρεσβύτες, οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες να έχουν την ίδια δυνατότητα, να έχουν πρόσβαση στην κοινωνία την ψηφιακή και να εποφελούνται και να χρησιμοποιούν αυτήν. Και γι' αυτό συμβαίνει το εξή. Έχουμε ως στόχο φυσικά όλοι, όλοι οι θεσμοί να έχουν αντίστοιχες ιστοσελίδες που με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούν, αλλά υπάρχει επιθυμία και εξακολουθούμε να την έχουμε αυτήν, ώστε για εκείνους τους θεσμούς και όργανα που πραγματικά για τις μικρο μικροεπιχειρήσεις, τις πιο μικρές δηλαδή επιχειρήσεις θα πρέπει να ανεβρίσκουν λύσεις που να μπορούν να προσανατολίζονται και υπό τις αρχές εκείνες που πάντα εσείς σε αυτόν τον τελευταίο καιρό πρόεδρε προσπαθήσατε να προαγάγετε να μην επιβαρύνονται δηλαδή αυτές ε, οι επιχειρήσεις υπέρμετρα. Σε κάποιες χώρες υπήρξαν δυσκολίες ε, για τη δραστηριότητα, αντιμετώπισαν δυσκολίες ε, οι μικροεπιχειρήσεις και πιστεύω ότι αυτό τώρα θα μπορεί να είναι μια μεσαία οδός βιώσιμη, μια μέση οδός βιώσιμη που θα μπορέσει να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων να μπορέσουν να ανταγωνιστούν και να επιβιώσουν. Το πεδίο εφαρμογής, αλλά ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο συνάδελφος, το κατέστησε ήδη σαφές, βήμα προς βήμα διευρύνεται σταδιακά από το Ευρωκοινοβούλιο προς όλες αυτές τις πτυχές και συνιστώσεις. Για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να πετύχουμε τις, μικροεπιχειρήσεις ε, να μπορέσουμε ξεχωριστά να τις αντιμετωπίσουμε. Και το πρόβλημα που έχει ο κύριος Στρασκόφσκι στην Πολωνία, οι μικρο, μικροεπιχειρήσεις ε, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με την, τις που έχουν, ώστε ξεχωριστά να υπάρξουν ρυθμίσεις για αυτές από τα κράτη-μέλη όπως γίνεται ήδη από, τα, ε, από τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Υποστηρίζει αυτή τη σταδιακή προσέγγιση ο κύριος Στρασκόφσκι ώστε ε, κατά την αρχή του 2015 να ξεκινήσουμε και το 2017 όλες οι επιχειρήσεις να εντάσσονται σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να μπορέσουν να έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν έτσι ώστε κυρίως το live audio content να προχωρήσει, να μπορέσουμε δηλαδή σε σχέση με αυτό το εγχείρημα να σημειώσουμε πρόοδο. Εκφράζει την ικανοποίησή του ο κ. Στρασκόφσκι ότι μια ομόθυμη προσέγγιση είναι αναγκαία ώστε κινητή τι η κινητή δράση ε, μέσα σε ευέλικτα πλαίσια να μπορέσει να λειτουργήσει. Να μπορέσουν όλα αυτά να οδηγηθούν σε μια ενιαία εφαρμογή ώστε ε, ο εξοπλισμός ε, ε, και η διαμόρφωση να προβλεφθούν και να εκτελεστούν όπως προβλέπονται από αυτήν την οδηγία. Είμαι βέβαιος ότι ως Υπουργός μπορεί να μεριμνήσει να επιτεθούν αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας του και έτσι λοιπόν να ευελπιστώ ότι ομόθυμα θα εγκρίνουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Good. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πέρεθ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος του συναδέλφου για το έργο που επιτελέστηκε και για τη συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές. Αυτή η οδηγία είναι αναγκαία και σκόπιμη για να δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες και τα αιτήματα των πολιτών που διεκδικούν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα και τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι τα ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πρεσβύτες που ζητούν να δοθούν λύσεις στις ανάγκες ανάγκες τους και να πάψουν να υπάρχουν προσκόμματα και εμπόδια. Η ομάδα μου εκφράζει την ικανοποίηση της ε, για το έργο που επιτελέστηκε και για τις 30 συμβιβαστικέ τροπολογίες. Θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, το δυνατόν στο μεγαλύτερο βαθμό και θεωρώ ότι, το, ότι συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα μεγάλο μέρος αυτών είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για μας οι τελικοί χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες και ιστοπύλες στο διαδίκτυο όλων των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Και οποιαδήποτε κινητή ε, δυνατότητα ως εξοπλισμός ε, να μπορεί να ε, έχει τη δυνατότητα σε ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής για να είναι προσβάσιμες οι νέες τεχνολογίες από τους πολίτες και νέες δυνατότητες. Απευθύνω έκκληση και ότι η έγκριση αυτής της οδηγίας σταδιακά θα μπορέσει να επιτευχθεί το νωρίτερο δυνατόν. Ξεκινά ήδη από το 2015 και μέχρι το 2017 όλες οι επίσημες δημόσιες ιστοσελίδες και ιστοπύλες, κρατικές αλλά και ιδιωτικές αλλά δημόσιου χαρακτήρα να μπορούν να είναι προσπελάσιμες, να είναι προσβάσιμες για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έγκστρομ. Συγγνώμη, είχα χάσει τον κατάλογό μου. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής και οι προλαλήσαντες σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί όλο και περισσότερη συνένεση έχουμε ως προς αυτό το θέμα και αυτό πραγματικό είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι ήταν αρκετά στενή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή, αλλά άκουσε διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεύρυνε κάπως το πεδίο εφαρμογής. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή και η έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους σας και θα περιμένω με αγωνία την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ χαίρομαι που επιτέλους ε, καταλήξαμε στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, θα τις υποστηρίξει όλες η ομάδα μας. Είναι πραγματικά ενημερωμένες. Δεν θέλαμε να είναι παροχημένες πριν καν αρχίσει να ισχύει ε, η λύση που προτείνουμε. Θέλουμε τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις. Εμείς θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κλπ. Οπότε χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που υπάρχει η τροπολογία 17 που μιλάμε για το περιεχόμενο ιστοτόπων και την ευθυγράμμιση του με την οδηγία. Όπως επίσης και τη συμβιβαστική 5 που μιλά για το πεδίο εφαρμογής ε, του εγγράφου. Είναι πολύ σημαντικό οι ιστότοποι των δημοσίων οργανισμών να καλύπτονται, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε και στους τόπους των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει κάποια από τα καθήκοντα των δημοσίων οργανισμών. Να συγχαρώ λοιπόν τον εισηγητή για το διορισμό του στην πολωνική κυβέρνηση και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να κάνετε λόμπι στον κύριο Τσασκόφσκι εκ μέρους μας, κάτι το οποίο είναι καλό. Η κυρία Στάιλερ, θέλει κανείς άλλος μετά την κυρία Στάιλερ να πάρει το λόγο. Όχι, ωραία. Κυρία Στάιλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τσασκόφσκι για την ε, ε, μετάβασή του στην Πολωνία ε, ως Υπουργού. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στην πολωνική κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει για την προώθηση των ε, θεμάτων που έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε, αλλά και μελλοντικών θεμάτων. Όταν συμβαίνει αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους πάντοτε να έχουν επαφή με την Επιτροπή μας. Συνήθως το κάνουν και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όσον αφορά τώρα ε, την έκθεση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή γιατί έλαβε υπόψη και δικές μου τροπολογίες τις συμβαστικές και δεν είναι εύκολο αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν για τη συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να υπάρξει κάποια λογική συμφωνία για το θέμα αυτό πριν τη διακοπή ενόψη των ευρωεκλογών γιατί κάποια από αυτά που έχουμε επιτύχει, ε, γιατί αυτό είναι μεταξύ των πραγμάτων που έχουμε επιτύχει και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εν ώψη των ευρωεκλογών. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ό,τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να προωθήσουμε τη διαδικασία ώστε κάτι ιστότοποι, κάποιοι ιστότοποι που δεν έχουν ευθυγραμμιστεί ακόμη να ευθυγραμμιστούν να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά ξανά και με την Ελληνική Προεδρία, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, ε, θα το δούμε στις αρχές Ιανουαρίου. Ήταν πολύ καλή λοιπόν η συνεργασία μας. Περιμένω εναγωνίως την αυριανή ψηφοφορία. Ελπίζω ότι στο τέλος ε, θα, είναι πολύ επωφελέ αυτό που θα προκύψει για όλους όσους δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση στους ιστοτόπους των δημοσίων οργανισμών. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ο, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Ζαματά είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας και να σα δώσω το λόγο να, να σχολιάσετε συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρώ για τις προσπάθειές σας. Προφανώς η Επιτροπή σας έχει μια πολύ καλή κατανόηση ενός πολύ δύσκολου θέματος και πολύ περίπλοκου. Ο στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι να είναι κατάλληλη πρόταση για το στόχο που θέλει να επιτύχει. Θέλουμε να ε, αξιολογήσουμε όλες τις συνέπειες, ειδικότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες σχετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εξίσου αποτελεσματικά και επικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρξει συνένεση κατά τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις της τρέχουσης, ελπίζουμε ότι και εκείνες θα συμβάλλουν. Ελπίζουμε ότι μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα έχει εγκριθεί το κείμενο ώστε να υπάρξει απλοποίηση ορισμένων άρθρων και επίσης επίζουμε να υπάρξει ε, επιτυχές κλείσιμο του θέματος αυτού ε, εντός της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χατζημαρκάκης, θα θέλατε παρακαλώ να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο τελευταίο θέμα. Να απαντήσω όμως, συγγνώμη πρώτα, στον κύριο Σβάπ για τις, μικρομεσές, για τις μικρές επιχειρήσεις. Πράγματι, τες αντιμετωπίζουν προβλήματα και όλες οι βέβαια επηρεάζονται οι επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο. Το θέμα είναι να υπάρχει σωστή μεταχείριση και δίκαιη μεταχείριση. Γι' αυτά που είπα ο κύριος ε, Μπίλαντ ε, για, τις, ε, για τα κινητά εμείς ε, ε, μένουμε στο θέμα των ε, υπηρεσιών από πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών ή καλύτερα των υπηρεσιών που παρέχονται από, από φορείς του δημοσίου. Φυσικά το να εκτιμήσουν Σκανδιναβοί την προσπάθεια που ε, έχει γίνει, ιδιαίτερα από τον κύριο Έγκστρομ, είναι πάρα πολύ θετικό για μένα. Πράγματι υπήρξε μια λογική από πλευράς της δικής μας ομάδας έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας το σκανδιναβικό υπόδειγμα έχει μεγάλη σημασία η εκλογής να μπορέσει έστω και να εγκρίνει μια τέτοια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πόσο μάλλον να την βελτιώσει και να κάνει κάτι θετικό για την κοινωνία, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση. Η ελληνική προεδρία έχει προετοιμαστεί σωστά. Οι επαφές που ε, είχαμε μέχρι τώρα μου έδειξαν ότι γνωρίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις λεπτομέρειες. Μου έδωσαν και κάποια επιπλέον στοιχεία για το τι πιστεύουν ε, οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι λέγουν ότι περιμένουν το ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς, το οποίο θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο, αλλά αν περιμένουμε τον Φεβρουάριο αυτό σημαίνει ότι η παρούσα πρόταση δεν θα ολοκληρωθεί. Γιατί υπάρχει και μια διαδικασία, θα έλεγα, ψήξης, η οποία δεν θα έχει δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν τυχόν πάμε τον Φεβρουάριο. και είμαι ευγνώμων προς την Ελληνική Προεδρία που μου υπενθύμησε αυτές τις λεπτομέρειες και μου έδειξε ότι είναι δυνατόν κάποιες επιμέρους προτάσεις ακόμα και τώρα να γίνουν δεκτές στις συμβιβαστικές. Λοιπόν, είναι εύκολος ο στόχος, ας τον πετύχουμε. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά δραστήρια δουλειά σας. Είχαμε οργανώσει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για τα θέματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό γιατί πάρα πολλοί θίγονται γύρω από τα θέματα αυτά. Ελπίζω να υπάρξει σημαντική πρόοδος. Σας ευχαριστώ που κάνατε και τις προκαταρκτικές αυτές επαφές με την Ελληνική Προεδρία. Θα ψηφίσουμε το θέμα αύριο. Από ό,τι φαίνεται θα υποστηριχθούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες και θα σας δώσουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά θα τα πείτε αυτά με τους κοιόδης. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε ένα νέο θέμα, ένα από τα τελευταία νέα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε, η έκθεση Μπίλαν, που είναι γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ ουσιαστικά για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ενιαία αγορά, για την ψηφιακή μάλιστα αγορά, όπου οι πληρωμές με ηλεκτρονικές κάρτες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι οι προμήθειες, οι διατραπεζικές προμήθειες στις συναλλαγές με κάρτες. Ε, έχουμε και τον κύριο Μπόρισοφ, ο οποίος παρακολούθησε ένα τμήμα της συζήτηση σήμερα και ο οποίος είναι σκιώδης για το ΕΛΚ. Έχουμε την εκπρόσωπο την κυρία Βερνιό από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, ο κύριος Ένστρομ για τους Πρασίνους, όχι δεν ξέρω αν ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, ε, ή θα περιμένουμε κάποιον άλλον από τη φιλελεύθερη ομάδα. Κύριε Χατζημαρκάκη, είστε σκιώδης για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, λέει ο κύριος Χατζημαρκάκης. Θα δώσω καταρχάς τον λόγο στον κύριο Μπίλαν. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Οπότε δεν θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη επιπτώσεων λοιπόν. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, κανονικά θα έπρεπε να παρουσιάσει την μελέτη επιπτώσεων για την πρόταση του κύριου Μπίλαν. Δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν φτάνει τώρα. Εν πάση περιπτώσει δύο λεπτά νωρίτερα είμαστε μόνο. Ας πάρει το λόγο ο κύριος Μπίλαν για να παρουσιάσει το θέμα του αμέσως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, οι διαπραγματεύσεις από πλευρά του Συμβουλίου έχουν κύρια σημασία για την λειτουργία της οικονομίας. Ταχεία καινοτόμα και ε, πολύ ε, ε, λιγότερο δαπανηρές οι συναλλαγές αυτές από τις ε, συναλλαγές σε μέτρητα. Ένα ωστόσο από τα στοιχεία ήταν το, για την ανάπτυξη ενιαίας εσωτερικής αγοράς το εγχείρημα των τεσσάρων ε, στοιχείων. Δηλαδή πολυμερών κειμενόμενων τελών. Πολλές φορές ε, οι χρήστες δεν γνωρίζουν ε, την ύπαρξη αυτών των τελών και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δυνατότητα ε, για τους επιχειρηματίες να βρεθούν οι αναγκαίες δυνατότητες. Οι δυνατότητες χρήσης καρτών συνεπάγεται πολλές φορές και η τέλη. Αυτό το οποίο προτείνεται εδώ με άλλα λόγια είναι ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας συναλλαγές εσωτερικής αγοράς ε, πληρωμών στις συναλλαγές. Ταυτοποίησε, εντόπισε έναν αριθμό προσκομμάτων και εμποδίων εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει κάποια ε, βήματα και διαβήματα για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τούτων λεχθέντων, η έγκριση ε, των στοιχείων αυτών των οροσίμων για τα τέλη είναι ένα μείζον βήμα για την βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η υλοποίηση των, των τεσσάρων ελευθεριών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα επικεντρωνόμενοι εστιαζόμενοι στους ίδιους τους καταναλωτές Πιστεύουμε ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα εναλλασσόμενα τέλη όσον αφορά εσωτερικές και εσωτερικές ε, συναλλαγές ε, και συγκυρίες αποφάσισα να μην υπάρξει όμως παρέμβαση στα όρια των ΚΑΠΣ διότι θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πλέον Στου κόλπου τη δικής μα κοινοβουλευτική Επιτροπής θα μα δώσει τη δυνατότητα να προαγάγουμε μια καλύτερη ε, λύση. Προβληματιζόμενοι για αυτές τις ρυθμίσει, πρέπει να προβληματιστούμε και για την επιβολή προστήμων ή κυρώσεων για να μην υπάρξει παράκαμψη ή αποφυγή ε, συμμόρφωσης με αυτές τις ε, διατάξεις. Πρέπει επίσης να είμαστε αμερόληπτοι ε, όσον αφορά την ημερήσια διάταξή μας σε σχέση με τα θέματα αυτά. Επίσης θα πρέπει τα τέλη αυτά να προσαρμόζονται ανάλογα με αυτές τις ανάγκες των ηλεκτρονικών ψηφιακών συναλλαγών σε σχέση με τη χρήση για παράδειγμα καρτών ε, έναντι της χρήσης ε, καρτών καταναλωτών. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να διαγραφούν, να αρθούν ε, οι διατάξεις όσον αφορά τις εμπορικές κάρτες. Δεν βρίσκω να υπάρχουν επαρκείς λόγοι. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ξεχωριστές διατάξεις. Επίσης, για τον ορισμό της κάρτας πληρωμής στο άρθρο 2 αυτή η αγορά μεταβάλλεται η μεταχείς ρυθμούς, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Θα πρότεινα λοιπόν να υπάρχει μικρότερη συντετμημένη περίοδος αναθεώρησης ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να επανεξετάσει και ταχύτερα να αναθεωρήσει αυτές τις διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ε, πρόσφατες εξελίξεις ε, σε αυτή την αγορά και τις πρακτικές ε, που ακολουθούνται από πλευρά των συναλλασσομένων. Επίσης έχουμε και την πρόταση να συνμηθεί η περίοδος για την αναθεώρηση διότι πιστεύουμε ότι διετής περίοδος ε, είναι υπερβολικά μακρά για την, ε, τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν σε σχέση με τις διασυνοριακές συναλλαγές. Σε πολλές χώρες τέτοιου είδους ε, διατάξεις ήδη λειτουργούν σήμερα. Αυτές οι διαμορφωμένες και διαφοροποιημένες περίοδοι μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό ε, όσον αφορά την αγορά καρτών πληρωμών. Το άρθρο 6 καταργεί οποιαδήποτε εδαφικά όρια ε, σε σχέση με την έναρξη λειτουργίας αυτών των, ε, σε ισχύ αυτών των διατάξεων και πρέπει σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο να δούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία σε επίπτωση για την λειτουργία της αγοράς. Για το άρθρο 7, προσωρινή προσωρινός αποκλεισμός, ε, εξαίρεση από αυτό το άρθρο νέων καρτών ή νέων συστημάτων, καθώς θέλουμε να προαγάγουμε την ε, λειτουργία, των, την χρήση των καρτών, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ε, υπερβάλλουμε με την επιβολή περιοριστικών διατάξεων ή περιορισμών, διότι πρέπει να μεριμνήσουμε να εμπλακούν και να συμμετάσχουν στην αγορά το δυνατόν περισσότεροι. Τώρα, από πλευρά των κρατών μελών για να μπορέσει να ε, δημιουργηθεί, να αποκτηθεί μια συνολική σφαιρική εικόνα του πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα στην αγορά και να μπορέσουν να ακολουθηθούν, να υιοθετηθούν οι βέλτιστες ε, δράσεις για να επιληθούν τα προβλήματα. Με ιδιαίτερη χαρά προσβλέπω στο να ακούσω τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας συνάδελφοι σε μια καρποφόρα συζήτηση. well, Νομίζω ότι ήρθαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εκπρόσωπος να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για την αξιολόγηση, τη μελέτη επιπτώσεων. Ίσως όμως εφόσον και άλλοι συνάδελφοι πρέπει να πάρουν το λόγο, καλύτερα να δώσω πρώτα το λόγο σε εκείνους και να σας δώσω το λόγο μετά. Ο κύριος Μπόρισοφ ε, από το ΕΛΚ και η κυρία Στάιλερ είναι εδώ επίσης. Η κυρία Βερνιόχη, η κυρία Στάιλερ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κύριε Μπορισόφ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη, όπω επίση και τον εισηγητή, τον κύριο Μπίλαν. Ε, χρειάζονται πράγματι μια ολοκληρωμένη αγορά πληρωμών ε, οι πολίτε, οπότε συμφωνώ με το στόχο τη πρόταση. Όμω το πρόβλημα των προμηθειών είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσέξουμε τον αντίκτυπο των ενδεχομένων αλλαγών. Να επικεντρωθώ λοιπόν στα εξή ζητήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτον, τα ανώτατα όρια των διατραμετών τραπεζικών προμηθειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σε διασυνοριακό και εθνικό επίπεδο ένα 0,5% για τη χρήση των πιστοτικών καρτών, ε, κάτι το οποίο θα μειώσει βεβαίως ε, τα τέλη και θα μειώσει και τις τιμές των υπηρεσιών αυτών για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι, το, οι τιμές αυτές βασίζονται σε μια αξιολόγηση των τιμών ε, ανάλογα με, το κατά ανάλογα με τη διαφορά που θα υπήρχε αν είχαν πληρωθεί μετρητής αυτά τα ποσά ή με κάρτες. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, ε, οι πληρωμές μέσω καρτών ε, είναι πολύ ανεπτυγμένες και είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές από ό,τι σε άλλες χώρες, άρα θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με τις πληρωμές μέσω το ανώτατο όριο των προμηθειών, αν ήταν ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν θα ε, αντανακλούσε σωστά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα καλό στην Πολωνία, για παράδειγμα, έχουμε την αντίθετη κατάσταση. Θα χρειαζόταν επιπλέον επένδυση για να υπάρχουν υποδομές πληρωμών μέσω καρτών κάτι το οποίο καλύπτεται από τις διατραπεζικές προμήθειες, διαφορετικά θα έπρεπε να αυξηθούν τα τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες στους καταναλωτές και ο καταναλωτής θα πλήρωνε την ύφη. Οπότε ε, πρέπει να δούμε και τις νέες τεχνολογίες, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Μπορούμε να σκεφτούμε τη λύση, για παράδειγμα, ένα μέσο όρο, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τις διάφορες αγορές πληρωμών καρτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το διασυνοριακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα μπορούσε να διαλέξει μια τράπεζα εκτός της χώρας του, που θα προτείνει καλύτερα τέλη. επομένως χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα θα σήμαινε χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες γενικότερα. Η τρέχουσα πρόταση δημιουργεί μία ρυθμιζόμενη και μη ρυθμιζόμενη περιοχή κάποιες ε, κάρτες όπως οι πιστοτικές κάρτες ε, την χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τις εμπορικές κάρτες. Όμως αυτές δημιουργούν τα περισσότερα τέλη για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο ε, στο θέμα αυτό και να αξιολογήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο στους καταναλωτές. υπάρχει ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τον καταναλωτή ότι όλες οι κάρτες πρέπει να γίνονται αποδεκτές ανεξαρτήτως τόπου έκδοσης τους. Αν κάποιος έχει ας πούμε ένα, μια Visa ή μια Mastercard ε, πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει αποδεκτή. Η πρόταση ε, του άρθρου 10 αλλάζει κάπως τα πράγματα και αφορά μόνο τις κάρτες, ε, τις ε, χρεωστικές για παράδειγμα, ε, που θα ρυθμίζονται συνολικά να έχουν τις ίδιες τιμές. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε καλύτερα το θέμα αυτό, γιατί ο αντίκτυπος θα είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορισόφ, λέει πρόεδρος, η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα <clears throat> να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτέλους θέλει να θέσει ένα τέλος ε, στα τόσο σκοτεινά αυτά θέματα των διατραπεζικών προμηθειών. Θα ήθελα να διαβρύνω το θέμα όχι μόνο στις πληρωμές τις, ε, με κάρτες, αλλά και τις αναλήψεις, τις ηλεκτρονικές κτλ. Το θέμα Λοιπόν, το θέμα σε καμία περίπτωση δεν είναι να αμφισβητήσουμε ε, την ύπαρξη αυτών των προμηθείων, αλλά μερικές φορές ε, η προμήθεια αυτή, το μέγεθός τους είναι πολύ υψηλό, ποικίλει πάρα πολύ από μια χώρα στην άλλη, από μια κάρτα στην άλλη και αυτό είναι μια τροχοπέδη στο εμπόριο και ένα πραγματικό φράγμα ανάμεσα στις εθνικές αγορές πληρωμών. Είναι πρόβλημα για τους εμπόρους και φυσικά για τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ολιγοπόλια. Χαίρομαι λοιπόν με τον εισηγητή που υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πληρωμών. Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες και τους δισταγμούς που υπάρχουν ακόμα και εδώ στο Βέλγιο για πληρωμές με κάρτες. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή πρόθεση των εμπόρων που ορισμένοι προτιμούν τις πληρωμές μετρητά αλλά λόγω των υψηλών προμηθειών των τραπεζών που οδηγούν μερικές φορές ε, στην αύξηση της τιμής της πληρωμής με κάρτας και στο να μην προτείνεται η πληρωμή με κάρτα για μικρά ποσά. Σχετικά με τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπίλαν τον ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαιτέρως ε, την προσπάθεια την οποία κάνει για να διευκρινίσει το τι εννοείται ε, κάρτα πληρωμών, τι σημαίνει κάρτα πληρωμών και η πρόθεσή του είναι πάρα πολύ καλή για την διαδικασία εφαρμογής των τοπικών ρυθμίσεων, γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ρυθμίσεις, σε άλλες όχι. Μέχρι τη στιγμή που θα καταθέσουμε και τις τροπολογίες θα κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις προς τον εισηγητή. Έχουμε όμως όλοι την ίδια επιθυμία να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση υπέρ των εμπόρων, υπέρ των καταναλωτών και να πάψει πλέον αυτή η διάσπαση, η ουσιαστική διάσπαση της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος σκιώδης που θα ήθελε το λόγο η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και τον εισηγητή και τους σκιώδης. Εμείς ε, ε, έχουμε γνωμοδότηση εδώ. Υπάρχει ενισχυμένη όμως συνεργασία. Όχι, απλά ήθελα αυτή τη διευκρίνηση. Κρίμα είναι, γιατί ε, φαίνεται ότι υπάρχει χώρος εδώ για να συνεισφέρουμε και με διαφορετικό τρόπο. Το θέμα της διαφάνειας είναι νομίζω βασικό στα πλαίσια της συγκεκριμένης συζήτησης. Και εγώ όπως και πολλοί άλλοι ε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ενήμερη για τέτοια θέματα, αλλά σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω και κατάλαβα πώς λειτουργεί το σύστημα και κατάλαβα πώς προχωρά το σύστημα ε, με ξεκάθαρο τρόπο και γι' αυτό και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση γιατί η διαφάνεια εδώ δεν υπάρχει ουσιαστικά και θα πρέπει το σύστημα να καταστεί πολύ πιο διαφανές και για τις επιχειρήσεις και για τους πελάτες. Η συζήτηση αφορά το να είμαστε διαφανείς, δίκαιοι και να κατανοήσουμε τα προβλήματα καλύτερα. Ταυτόχρονα όμως οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις κάρτες αυτές θα πρέπει να προστατεύονται από απάτες και καταχρήσεις και θα πρέπει να δίδουν εγγυήσεις σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν μέχρι τώρα τις κάρτες ηλεκτρονικές πληρωμών όπως Visa, Mastercard κτλ. Βλέπουμε ότι σε διάφορες χώρες υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Ο κύριος Μπίλαντ αναφέρθηκε σαν παράδειγμα στο τι ισχύει στην Πολωνία, το τι ισχύει στη Γαλλία, το τι ισχύει κάθε φορά σε διαφορετικές χώρες. Το θέμα είναι ε, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες λειτουργούν με διαφάνεια, κάποιες άλλες όχι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα παραδείγματα αυτά σαν βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχει και το θέμα του κόστους προς τους καταναλωτές. Αν τυχόν, σαν παράδειγμα σύμφωνα με τις στατιστικές, το κόστος εφαρμογής του συστήματος στον καταναλωτή που χρησιμοποιεί τη Visa θα είναι 35 λίρες το μήνα, μου είπαν. Δεν ξέρω τι είναι αυτές οι δηλώσεις, αν είναι αληθείς μπορεί να μας διαβεβαιώσει η Επιτροπή ότι δεν θα επιβαρύνουν όλα αυτά τον πολίτη. Και όταν αναφέρομαι σε κάποιες μικρές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών γιατί έχουν υψηλό κόστος. Πρέπει το κόστος και συγκεκριμένα η προμήθεια να οριστεί με σωστό τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργήσει προβλήματα ε, ούτε στους εμπόρους αλλά ούτε και σε μια χώρα σαν παράδειγμα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις σχετικά με το κόστος προς τον ε, ε, καταναλωτή που πληρώνει ο καταναλωτής. Αν υπάρξει ευρωπαϊκό σύστημα ε, οι προμήθειες αυτές θα αυξηθούν ή θα μειωθούν. Και το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται αναχώρα πώς κρίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ θα ήθελα να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που απαιτούν οι έμποροι και σε αυτά τα οποία χρειάζεται ο πελάτης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσπάθειά σας. Είναι ένας τομέας στον οποίο όταν αρχίζει κανείς να εξετάζει προσεκτικά ανακαλύπτει ότι απαιτούνται πάρα πολλές παρεμβάσεις και λύσεις και ελπίζω οι λύσεις αυτές να έρθουν το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα που ελέγχθησαν. Κάνοντας λόγο για αυτά τα θέματα μιλάμε για διαφάνεια, κατά του κερματισμού της αγοράς. Δεν έχουμε διαφάνεια. Ο κύριος Μπίελαν το είπε. Είπε ότι οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τι πληρώνουν όταν χρησιμοποιούν τέτοιες κάρτες. Ποτέ δεν ξέρουν θα έλεγα. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι και κρυμμένα, ε, κόστη, συγκαλυμμένα τέλη αυτά και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει για να έχουν μια επιλογή και να συνειδητοποιήσουν το τι συμβαίνει οι πολίτες και τι πληρώνουν με τέτοια τέλη. Όλοι υφιστάμεθα τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης σε σχέση με καταστήματα, μαγαζιά, κάποιοι δεν χρησιμοποιούν, δεν δέχονται τέτοιες κάρτες ή λένε σήμερα δεν λειτουργεί τούτο ή το άλλο και δεν μπορεί να γίνει δεκτή η κάρτα σας κτλ. Θέλουν μετρητά διότι θέλουν να εξοικονομήσουν αυτά τα κόστη, αυτά τα τέλη. Φυσικά επίσης θα ήθελα οι περισσότεροι, όπως και οι περισσότεροι από εμά, να μην υπάρξουν ρυθμίσεις και υπερβολικές ρυθμίσεις. Υπάρχει όμως ήδη μία απειλή επιβολής τέτοιων τελών. Ίσως ε, η λύση μπορεί να επιτευχθεί πριν από τέτοια επιλογή. Εγώ πάντα επιλέγω να μην υπάρξουν διατάξεις και ρυθμιστικές τέτοιες ε, ε, επιβολές διατάξεων. Ωστόσο όμως ίσως μπορεί να βοηθήσει η απειλή τέτοιας επιβολής διάταξης να επιληθεί το πρόβλημα. Υποστηρίζω την πρόταση επίσης του του κυρίου Μπιέλλαν να συνμηθούν οι περίοδοι, μεταβατικές περίοδοι. Γιατί να περιμένουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Well, thank Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό τον πρώτο γύρο. Αυτό που κάναμε προηγούμενα σε σχέση με τις προτάσεις, είχαμε μελέτη επιπτώσεων μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έκθεση του εισηγητή. Τώρα έχουμε μια αντιστροφή των όρων. Καλό θα ήταν τώρα να δίναμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να μας πληροφορήσει τι έγινε. Ε, δυστυχώς δεν είχαμε τα στοιχεία σας ε, και τις διαφάνειες ε, και έτσι δεν μπόρεσαν να δειχθούν. Ίσως ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν ιστερότερα να μας γνωστοποιηθούν και σε σχέση και με τα στοιχεία που γραπτά μπορούν να διατεθούν. Λοιπόν, αναμένουμε να ακούσουμε από πλευρά σας έχουμε αυτή τη συνεδρίαση, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12.30 αν χρειαστεί από πλευρά σας. Υπάρχει πολύς χρόνος, επαρκής χρόνος για τη συζήτηση, σας δίνουμε το λόγο και σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίασή μας. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που προσέρχεστε σε μια τέτοια συνεδρίαση και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, είναι που αφοράτε σε σχέση με αυτό το θέμα, διότι συζητώνται πολλά θέματα σε σχέση με τα όσα βρίσκονται υπό εξέλιξη και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι δικές σας αντιδράσεις. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε και τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς ε, συν συντάκτη στην εκπόνηση αυτής της ε, πρότασης. Ε, πολύ θετικό αυτό. Ναι, πράγματι, έντονα συνεργαστήκαμε σε βάθος σε αυτό το πακέτο μέτρων για την ρύθμιση για τα αναλασσόμενα τέλη και την οδηγία ε, αυτά τα τέλη θα συζητήσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Επενούμε για το σχέδιο έκθεσης, επένους θέλουμε να εκφράσουμε. Πράγματι ζητούμε συγγνώμη, διότι διότι δεν υπήρχε εξοικείωση σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου στη γενική μας διεύθυνση, δεν γνωρίζαμε ότι έπρεπε να σας γνωστοποιήσουμε ευθύς εξ αρχής τη δυνατότητα αυτή και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφανειών. Οι διαφάνειες σε σχέση και με τη μελέτη ε, επιπτώσεων που είχε ζητηθεί να συνταχθεί, δρατώμεθα τις ευκαιρίες της πρόσκλησης, πρόσκλησης ε, για να καλυφθούν τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε κάνουμε είναι για εκείνου που δεν έχουν εξοικειωθεί σε σχέση με τα εναλλασσόμενα τέλη, διακειμενόμενα τέλη, να σα δώσουμε μια επεξήγηση και να διευκρινίσουμε τι συμβαίνει με αυτά τα τέλη. Και αυτό το οποίο με τη μελέτη επιπτώσεων να επεξηγήσουμε κάποιε από τι επιλογέ που έγιναν στο σχέδιο ε, κανονισμού και να τοποθετηθούμε σε σχέση με κάποια ζητήματα και να ε, αντιμετωπίσουμε κάποιε παρανοήσει σε σχέση με το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο. Λοιπόν, για τα κειμενόμενα τέλη είναι πρώτα. Για εκείνους που δεν έχουν ε, γνωστό, ε, εξοικειωθεί με αυτά, τουλάχιστον όλοι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια θέματα χωρίς να τα γνωρίζουμε, να υπεξηγήσουμε όταν πάμε σε ένα μαγαζί και αγοράζουμε μια φωτογραφική μηχανή 100 ευρώ, εμείς ε, ως καταναλωτές θεωρούμε ότι δωρεάν γίνεται αυτό σε σχέση με τα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν για αυτή την πληρωμή. Θεωρούμε ότι δωρεάν χρησιμοποιείται η κάρτα μας. Όμως, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πληρώσει ένα ποσοστό στη δική του τράπεζα ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείτε. Και η τράπεζα θα πληρώσει 70% του ποσού αυτού που πληρώνει ο ιδιοκτήτης της τράπεζας στην τράπεζα που πηγαίνει στη δική μου τράπεζα. Έτσι έμεσα χρηματοδοτεί τη δική μου τράπεζα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για τη χρήση που, ε, της κάρτας που κάνω εγώ. Αυτή είναι η εναλλασσόμενη ε, κάρτα, το εναλλασσόμενο τέλος. Ε, και αυτά τα τέλη ε, εισπράττονται συλλογικά από τις διάφορες τράπεζες υπό την αιγίδα του ενός σφαιρικού συστήματος Mastercard ε, και άλλων συστημάτων. Οι τράπεζες ε, και στην πλευρά έκδοσης ε, και στην πλευρά ίσπραξής σα ε, συμφωνούν για τα ποσοστά τα οποία θα εισπράττονται και θα μετακυλίονται. Ποια είναι αυτά τα ποσοστά. Belgium Contact Card όταν τη χρησιμοποιώ εγώ θα είναι 5 cents για μια συναλλαγή 100 ευρώ. Αν χρησιμοποιήσω Mastercard κάρτα, ίσως όχι στο Βέλγιο αλλά σε μια άλλη ε, χώρα, τότε αν είναι μια πιστοτική κάρτα 10-20 cent για μια συναλλαγή. Διαφορετικά 70 ή 1-20. Αν χρησιμοποιήσω commercial card, εμπορική κάρτα που δίνεται από τον εργοδότη μου για ε, δαπάνες ε, αποστολών ε, ή εξόδων, τότε θα είναι ίσως 1,5 ευρώ ή 1,70. Και αν χρησιμοποιήσω American Express κάρτα που είναι ξεχωριστή, θα είναι γύρω στα 2,5 ευρώ ή ακόμα και 3 ευρώ αυτά τα τέλη. Όλες αυτές, όλα αυτά τα τέλη για την ίδια συναλλαγή και για την επιβάρυνση και του ίδιου του ιδιοκτήτη του καταστήματος για την αγορά. Η διαφορά είναι ότι σε σχέση με την ε, δική μου τράπεζα θα μου, δώσει κίνητρα να χρησιμοποιώ την πιο ακριβή κάρτα που δίνει μεγαλύτερα κέρδη για την τράπεζα. Θα έχω έτσι λοιπόν πρόταση με, με ανταπόδοση ταξιδίων, πόντων, μορίων ή άλλων ε, δώρων να χρησιμοποιήσω την πιο ακριβή μου κάρτα σε σχέση με κάποια άλλη. Είναι ένα σύστημα λοιπόν το, έχει, το οποίο συνεπάγεται μειονεκτήματα. Εμεί από πλευρά τη Γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα εδώ και πάνω από 20 χρόνια και με συνέπεια λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ τραπεζών είναι περιορισμό του ανταγωνισμού διότι αν συλλογικά συμφωνούν οι τράπεζες φόλων αυτών το κάνουν πολύ πιο δύσκολο για μια άλλη τράπεζα να συμφωνήσει και να διαπραγματευτεί για μια άλλη ξεχωριστή κάρτα με ξεχωριστά ε, τέλη. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο ε, με αυτή τη συλλογική συμφωνία τραπεζών καθορίζει κατόφλι ε, ή ανόφλια. Αν υπάρχει λοιπόν μια συλλογική συμφωνία να πληρώνονται 20 λεπτά, 0,20 ευρώ, αυτό θα είναι το κατόφλι κάτω από το οποίο ο έμπορος ποτέ δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Διότι οι εμπορικές τράπεζες θα γνωρίζουν ότι όλες οι άλλες τράπεζες θα έχουν συμφωνήσει για αυτό το ποσό. Αυτό είναι που αποκαλούμε περιορισμός του ανταγωνισμού. Και θεωρούμε ότι αν υπάρχει τέτοιος περιορισμός και είναι ανταγωνισμός, του ανταγωνισμού, απαγορεύεται αυτό από τους κανόνες και κανονισμούς για τον ανταγωνισμό. Εκτός αν υπάρχει εύλογη δικαιολόγηση. Και σε σχέση με τις τράπεζες αυτά που λένε είναι ότι είναι μια διμερή πολυμερής δίπλευρη αγορά και αυτό σημαίνει ότι μία πλευρά της αγοράς έχει μεγαλύτερο συμφέρον από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μέσα πληρωμών. Πολλές φορές έχουμε απέναντί μας τέτοιου είδους ε, ε, στοιχεία. Λένε ότι οι άντρες ε, έχουν, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον να πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο έναντι των γυναικών. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες πληρώνουν με κάρτες περισσότερο από ότι άντρες για παράδειγμα φιλοσοφία είναι αν ζητάμε από τους εμπόρους να πληρώσουν τότε οι κάρτες θα έχουν κίνητρα για την χρήση, για την χρήση τους. Θα έχουν προτερήματα αυτά για τους εμπόρους, θα είναι ασφαλείς, ε, ταχείες οι συναλλαγές. Εμείς ε, δεχόμαστε αυτό το πνεύμα αυτής της φιλοσοφίας αλλά δεν δεχόμαστε το ότι τα τέλη θα πρέπει να είναι τόσο υψηλά όσο είναι σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς την διαφορετική διαμόρφωση τελών σε σχέση με διαφορετικά κράτη πόσο μάλλον περισσότερο και μέσα στην ίδια, ε, σε μία και ίδια χώρα. Βλέπουμε λοιπόν για bank ε, ε, και οι άλλες κάρτες που πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τράπεζες ώστε να χρησιμοποιείται η κάρτα τους ευρύτερα. Το βλέπουμε αυτό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν καταργήθηκε το εθνικό πλαίσιο ξεκίνησε η Mastercard. Προσέφερε δύο λεπτά περισσότερα από ό,τι στο εθνικό πλαίσιο. Άρχισαν όλες οι τράπεζες να δίνουν Mastercard. Μετά ήρθε η Visa. Έδινε άλλα δύο λεπτά παραπάνω. Σε μικρή περίοδο πέρασαν στην ε, έκδοση εκδόσεων Visa καρτών οι τράπεζε. Δεν γνώριζαν όμω οι καταναλωτέ ότι το ποσοστό ίσπραξη αυξανόταν κατά δύο λεπτά περισσότερο για κάθε συναλλαγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μα ε, δημιουργεί δυσφορία όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμό να οδηγεί σε κεκριμένες ε, συγκαλυμμένε πληρωμέ από πλευρά τελών και αυτό να στρεβλώνει, να περιορίζει τον ανταγωνισμό κάτι που δεν δεχόμαστε. Υπό το πρίσμα των αρχών για τον ανταγωνισμό και υπό το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών. Επειδή οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι πληρώνουν έμεσα. Και όλα αυτά αυξάνουν τα τέλη και το κόστος υπηρεσιών και αγαθών. Και σε σχέση με την ε, American Express ε, οι άλλες κάρτες όλοι πληρώνουμε παραπάνω μέσω αυτής της ε, επιβολής τελών. Αν πληρώνω για παράδειγμα με μια φθηνότερη κάρτα ε, χρέωσης ε, πληρώνω και συνεισφέρω στην ε, χρηματοδότηση εκείνων που εκμεταλλεύονται, χρησιμοποιούν την έκδοση αυτών των καρτών. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι φτωχοί πληρώνουν υπέρ των πλουσίων και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε να γίνεται. Παρότι ασχολούμαστε με, την, με τα θέματα ανταγωνισμού εμπλέκονται και θέματα προστασίας των καταναλωτών σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι αυτά είναι τα, περι, τα ε, πιο πολλά προβλήματα και έχουν και σπουδαιότητα σε σχέση με την εμβέλειά τους τα τελευταία χρόνια. Και όταν κάνουμε λόγο για αυτά τα τέλη, η αναλογία των ε, τέλη είναι κάτι μεταξύ 10 έως 50%. Αν δει κανείς το λιανικό εμπόριο, σε κράτη-μέλη υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη πάνω από 60% τέτοιων συναλλαγών. Τώρα, αυτά τα θέματα έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και βάρος από ότι ε, όταν πληρώνει κανείς ε, μετρητά. Και έτσι αυτά τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα. Ερώτημα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την πρώτη εναλλαγή σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων. Είναι η μηδενική επιλεκτική λύση εναλλαγή. Να κάνουμε τίποτα δηλαδή. Το να κάνουμε τίποτα θα σημαίνει μηδενικό αποτέλεσμα. Δεν θα γίνει τίποτα. Έχουμε περιπτώσεις κατά της Mastercard και κατά της Visa. Προσφυγές δηλαδή. Και έχουμε καταλήξει και σε επιδιαιτησίες. Έχουμε και προσφυγή σε δικαστήριο για τη Mastercard αναμένουμε την ομολογία, την ε, απόφαση του 10 για αυτό το θέμα. Το αναμένεται κατά τα μέσα του επομένου έτους. Αφορά και μια απόφαση που υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε το 2007, όταν είπαμε ότι τέτοιου είδους ε, μετακυλιόμενα τέλη απαγορεύονται και δεν μπόρεσε να παρουσιάσει επαρκώς πιστικά επιχειρήματα η Mastercard κατά αυτής της τοποθέτησης. Είναι μια πολύ σύνθετη και περίπλοκη διαδικασία. Έχουμε ε, διεθνή πλαίσια τα οποία έχουν αναλάβει δεσμεύσει εναντί ημών να μειώσουν στο 0,2% ε, και 0,3% και πιο πρόσφατα η Βίζα προσέφερε και εκείνη το ίδιο να κατέβει στο 0,2-0,3% όσον αφορά ε, επιβολή τελών. Αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό αφορά τη Mastercard μόνο διασυνοριακές συναλλαγές για εκείνη και για τη βίζα τα τέλη για διασυνοριακές συναλλαγές. Όταν εγώ πάω στη Γαλλία για παράδειγμα και χρησιμοποιώ κάρτα βίζα μου εκεί, συν άλλα 10 κράτη-μέλη. Αλλά όχι τα πιο σημαντικά κράτη-μέλη για τις ε, συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τελών πάλι δεν θα μπορούν να αλλάξουν ή να ε, τροποποιηθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι το ίμιση των περιπτώσεων αυτών ε, αντιμετωπίζονται από τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές αρχές για τα θέματα ανταγωνισμού. Όμως, αυτό όμως θα πρέπει να δούμε σε σχέση με την επιτάχυνση και επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων τους περιορισμούς που θέτει. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι όλοι εργαζόμαστε σε σε διαφορετικά πλαίσια και περιπτώσει. Έχουμε διαφορετικέ καταστάσει στην Πολωνία και Ουγγαρία όπου υπάρχει μια απόφαση που βρίσκεται υπό έφεση. Υπάρχει άλλη απόφαση στη Γαλλία όσον αφορά για παράδειγμα την αρχή ανταγωνισμού. Έχουμε μια έναρξη διαδικασία που έχει παγώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε μια ολόκληρη σειρά κατακαιρματισμένων ε, ψηφίδων α το πω έτσι τη συνολική εικόνα. Θα υπάρξει ανάγκη να περάσει αρκετό χρόνο. μέχρι να συνδεθούν αυτές οι ψηφίδες σε μια συνολική εικόνα. Βλέπουμε ότι σχεδόν 90% των τελών σήμερα δεν εντάσσονται στα όρια τα οποία είχαν συμφωνηθεί σε σχέση με τη Visa και την Mastercard. Και αν δει κανείς τη συνολική εικόνα τώρα ε, σε σχέση με το 0,2-0,3 μπορεί να είναι χαμηλά τα τέλη. Λυπούμε που δεν έφερα τις διαφάνειες για να σας ε, ενημερώσουμε σχετικά. Αν δει κανείς τη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα τα τέλη για την Πολωνία, Ουγγαρία είναι καπλάσια από ότι αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πρόβλημα για την ενιαία εσωτερική αγορά. Εγώ, αν κάποιο που θέλει να προσφέρει κάτι καινούριο, μια κάρτα για την ευρωπαϊκή αγορά ή για πέντε κράτη-μέλη, αντιμετωπίζω το γεγονό ότι σε αυτά τα κράτη-μέλη οι τράπεζε ε, ε, αναμένουν να πληρώνω τα ίδια τέλη που πληρώνονται από τους άλλους που συμμετέχουν εκεί. Αυτό δημιουργεί διαφορές στα κράτη-μέλη και υπάρχει εδώ θέμα ανταγωνισμού και υπάρχει θέμα προσφυγής. Είναι παράνομα αυτά τα τέλη και δημιουργείται πρόβλημα αν θέλω εγώ να εισέλθω στην ευρωπαϊκή αγορά ως ανταγωνιστής. Και αυτό όχι μόνο εφαρμόζεται και ισχύει για ε, προγράμματα καρτών αλλά ισχύει και για προγράμματα διαδικτυακά και κινητές, δυνατότητες κινητών συναλλαγών με κινητές συσκευές Όλα αυτά τα συστήματα τα οποία εισάγονται ως καινοτόμα στοιχεία στην αγορά δημιουργούνται μείζωνα προβλήματα. Υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες και περιμένουν να πληρωθούν διαφορετικά τέλη οι τράπεζες σε διάφορα κράτη-μέλη. Και έτσι σε κάθε χώρα πρέπει να γνωρίζει κανείς ποιο είναι το μετακυλιόμενο κειμενόμενο τέλος για να γνωρίζουν τι θα ισχύει στο, να γνωρίζουμε τι θα ισχύει στο διαδίκτυο. Δεν είναι εύκολο αυτό και να διαφοροποιεί κανείς έτσι τα πράγματα για τα κράτη-μέλη και εδώ τίθεται θέμα λειτουργία τη εσωτερική αγορά που δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε. Αν ένα ε, λιανική εμπορία έμπορο θέλει να ε, κινηθεί και να χρησιμοποιήσει τα χαμηλότερα τέλη σε ένα γειτονικό κράτο μπορεί να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντα τι υπηρεσίε μια χώρα, μια τράπεζα για παράδειγμα στη Γερμανία για να ε, εξυπηρετηθεί. Όμω οι κανόνε του πλαισίου αυτού υποχρεώνουν την τράπεζα σε αυτή την περίπτωση να πληρώσουν το μετακυλιόμενο κειμενόμενο το τέλος σε σχέση με την τράπεζα της χώρας συναλλαγής. Μπορεί να πληρώνεται το τέλος που εφαρμόζεται μόνο στη χώρα εφαρμογής. Κάπου λοιπόν εδώ δεν λειτουργεί σωστά η ενιαία εσωτερική αγορά λόγω αυτών των διαφορετικών πλαισίων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια ενιαία λύση. Αυτά ουσιαστικά για τη μηδενική λύση. Να μην κάνουμε τίποτα αριθμιστικά που οδηγεί σε αυτή την κατάσταση όπως έχουμε σήμερα, που είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά με πολλά προβλήματα για όλους τους συναλλασσομένους. Να δούμε τι θα γίνει τώρα λοιπόν σε ευρωπαϊκή κλίμακα, διευκρινίζοντας προς τους καταναλωτές ποιο είναι το κόστος αυτών των πιθανών αλλαγών. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να ρυθμίσουμε κάποιο την κατάσταση. Καταρχάς, το, η πρώτη επιλογή είναι να ρυθμίσουμε μόνο τις διαμεθοριακές διατραπεζικές πληρωμές. Mastercard και Visa και τίποτα περισσότερο και ας προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε ρυθμίσεις έτσι ώστε οι έμποροι να μπορέσουν ε, να χαμηλώσουν και τις τιμές τους για τις ε, συναλλαγές τους. Να προτείνουμε δηλαδή στον κανονισμό αυτό ε, να είναι η πρώτη φάση αν θέλετε της εφαρμογής της πρότασης. Επαναλαμβάνω, πρώτη φάση φιλελευθερωποίηση όλων των διαμεθοριακών συναλλαγών ακόμα και αν πηγαίνουν οι πελάτες ε, ή οι έμποροι στο εξωτερικό και να γίνουν δεκτά τα ποσοστά των ε, διατραπεζικών προμηθειών που είναι αποδεκτά διεθνώς. Δεν αρκεί αυτό, γιατί ιδιαίτερα οι μικροί εμποροί θα μπορούν κεντρικά να χρησιμοποιούν μια τράπεζα για πάρα πολλές ε, χώρες. Από την άλλη οι μεγάλοι έμποροι θα ξεπερνούν τα προβλήματα σε διαφορετικές κλίμακες και να επενδύουν σε αυτές τις ε, ε, δυνατότητες. Αλλά αν είσαι ένα μικρό καπνοπολείο είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις εσύ διαφορετικά μέσα και να χρησιμοποιείς πολλαπλές διατραπεζικές υπηρεσίες. Η πρόταση λοιπόν αυτή του πρώτου σταδίου είναι καλή και θα μελτιώσει λίγο την κατάσταση, θα μειώσει λίγο το κόστος των προμηθειών, αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ισότιμος και δίκαιος τρόπος αντιμετώπισης ε, του προβλήματος από όλους. Ας θα μπορούσε να πει κανείς, ας αφήσουμε τα κράτη-μέλη να δούνε ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο της διατραπεζικής προμήθειας το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια διαμφισβήτητη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού. Από την άλλη, αν το κάνουμε αυτό, φιλελευθερωποιώντας τις διαμεθοδιακές συναλλαγές, ανοίγει στην πίσω πόρτα σε όλους τους εμπόρους λιανικής να διαφεύγουν. Αυτό λοιπόν σε μια πρώτη φάση είναι κάτι το καλό, αλλά δυστυχώς οι μικροί έμποροι είναι τα θύματα του συστήματος. Τελικά λοιπόν είναι αναπόφευκτο και θετικό τελικά για την εσωτερική αγορά να περάσουμε σε ένα ισότιμο πεδίο όπου και τα εσωτερικά τέλη των προμηθειών θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα διεθνή. Ποιο θα είναι αυτό το επίπεδο τώρα. Εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι το 0,2 και 0,3 που γίνονται δεκτά και από τα δύο σχήματα και από την ΒΙΖΑ για τις πιστοτικές κάρτες. Βλέπουμε ότι τα προγράμματα αυτά ε, βλέπουν ότι το ποσοστό αυτό λειτουργεί, ε, δεν έχουν καταρρεύσει αυτά τα σχήματα ε, και ευημερούν και αυξάνονται οι πωλήσει και οι συναλλαγές με πιστοτικές κάρτες. Αυτά. Νομίζω ότι έχω ήδη συμπεριλάβει και αρκετές άλλες δευτερεύουσες επιλογές στα πλαίσια της μελέτης επιπτώσεων. Τέθηκε ένα ερώτημα τι γίνεται με τα τριπλά σχήματα και εδώ απαιτούνται κάποιες εξηγήσει περαιτέρω. Το πρόβλημα που έχουν οι διατραπεζικές προμήθειες υπάρχουν γιατί οι έμποροι λιανικής έχουν την αδυναμία να αρνηθούν ορισμένες κάρτες ή να τις χρεώσουν περισσότερο. Και αυτές είναι οι λεγόμενες κάρτες ε, πίστοσης τις οποίες έχουμε πέρα από τις κανονικές πιστοτικές κάρτες. Αν δείτε τις κάρτες debit, σαν παράδειγμα, κατά μέσο όρο ένας Ευρωπαίος πολίτης έχει μια μισή τέτοια κάρτα και υπάρχουν ακόμα και παιδάκια και μωρά που έχουν τέτοιες κάρτες. Όλοι θα έχουμε τέτοιες κάρτες και θέλουμε να τις χρησιμοποιούν και ακόμα και αν οι προμήθειες είναι μερικές φορές υπερβολικά υψηλές για τους εμπόρους δεν μπορούν να τους αρνηθούν και δεν μπορούν και να τις υπερχρεώσουν γιατί θα πάνε σε άλλο λιανέμπορο. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι δύσκολο για τους εμπόρους λιανικής να ασκήσουν πιέσεις επί του ποσοστού προμήθειας. Γι' αυτό λοιπόν κάτι τέτοιο ε, θα μπορούσε ε, να επιληθεί σε σχέση με τις επιχειρηματικές κάρτες ε, εμπορικού τύπου που χορηγούν οι εργοδοσίες τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης. Η αμέξες σαν παράδειγμα που λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. Αυτές οι δύο κατηγορίες πιστοτικών καρτών έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς που είναι εύκολο για τον ε, πελάτη να πει ότι εγώ δέχομαι την debit και την credit που έχεις αλλά δεν δέχομαι την Amex. Ή και κάτι που θα μπορούσε να είναι πιθανό, δέχομαι την ε, ε, debit card που έχεις αλλά δεν δέχομαι την gold card που έχεις. Νομίζω λοιπόν ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο γιατί σε αυτή την περίπτωση ε, εμπλέκεται και ένα ενδιάμεσο επίπεδο που είναι ο εργοδότης ο οποίος ζητά την έκδοση της κάρτας για τους υπαλλήλους. Τίθεται το θέμα λοιπόν της διαφάνειας. Καταρχάς εδώ ε, θα πρέπει οι ε, έμποροι να γνωρίζουν το τι πληρώνουν για κάθε κάρτα οι τράπεζες μέχρι τώρα αναμειγνύουν τις προμήθειές τους, ενώ θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται για κάρτα τι ε, σημαίνει αυτό. Ο έμπορος πολλές φορές δεν ξέρει ακριβώς όταν πληρώνει ένα ποσοστό τι είναι αυτό το ποσοστό, δεν μπορεί να το αναλύσει. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο έμπορος λιανικής να έχει επιχειρήματα απέναντι στον πελάτη όταν αρνείται να χρησιμοποιήσει την κάρτα του πελάτη. Το ίδιο επίσης και με τις, ε, ε, ε, και με τις χρήσεις των κινητών τηλεφώνων που περνούν τα στοιχεία για τη χρήση των καρτών αυτών στο κινητό τηλέφωνο με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι πάντα ευδιάκριτος. Οι τράπεζες λοιπόν προφανώς θα ήθελαν να προωθήσουν τις πιο ακριβές κάρτες και να μην προωθήσουν τις φθηνότερες για τους πελάτες κάρτες. Το θέμα είναι να μπορεί να κάνει μία προεπιλογή ο έμπορος και να αποφασίζει ο πελάτης το τι θα χρησιμοποιήσει. Θα χρησιμοποιήσει. Αυτές είναι οι πιθανές επιλογές που έχουμε. Τέθηκαν και κάποιες ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε τρεις από τις ερωτήσεις σας. Uh, λοιπόν, η πραγματικότητα της αγοράς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες, όχι μόνο ε, ανάμεσα σε χώρες μέλη, αλλά και ανάμεσα σε τομείς. Αυτό που πληρώνετε για τη χρήση της κάρτας σας είναι διαφορετικό όταν πουλάτε αυτοκίνητα ή όταν ε, πουλάτε ε, ε, λιανική σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, προφανώς είναι διαφορετικά τα ποσοστά ποικίλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόστος χρήσης και το κόστος ε, έκδοσης, όχι και τόσο μεγάλες οι διαφορές, αλλά οι διαφορές αυτές ε, παραμένουν συνεχώς. Και να μην ξεχνάμε ότι οι διαφορετικές πραγματικότητες της αγοράς προκαλούνται και από τις προμήθειες. Σαν παράδειγμα είναι η Πολωνία και το ακούω αυτό πάρα πολύ συχνά. Στην Πολωνία υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι αυτές τις κάρτες, αλλά η Πολωνία μέχρι πολύ πρόσφατα, γιατί τώρα υιοθέτησαν κάποιες ρυθμίσεις, είχαν τις υψηλότερες προμήθειες στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια κάθε Πολωνός έχει μια κάρτα, αλλά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, γιατί μόνο στο 20% των εμπόρων ε, γίνεται δεκτές οι κάρτες αυτές. Οπότε χρησιμοποιούν την πιστοτική κάρτα για να πάνε σε, μια, ε, σε ένα, ε, σε ένα σημείο όπου ένα ATM παρέχει χρήμα να πάρουν το χρήμα και να πάνε να πληρώσουν με αυτό χρησιμοποιώντας την κάρτα τους πάντα. Λοιπόν, είναι ε, η κατάσταση διαφορετική. Εμείς θα θέλαμε οι έμποροι να δέχονται τις κάρτες πολύ περισσότερο. Η πολωνική κυβέρνηση δεν του εισάρεσε που είχε το υψηλότερο κόστος και τώρα έγιναν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μειωθεί. Υπάρχει πρόβλημα στην Πολωνία, υπάρχει πρόβλημα στην Ουγγαρία και στην Ιταλία αναμένεται νέα νομοθεσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των αγορών. Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα για τους καταναλωτές. ο φόβος ότι όπως έγραψαν κάποιες αγγλικές εφημερίδες θα χρεωθούν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα είναι αλήθεια Εξαρτάται πού τοποθετείται κανείς. Έχουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στην έκδοση για την έκδοση τη κάρτα του, Αυτό εξαρτάται από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα πιστοτικά ιδρύματα. Και είδαμε εντελώ διαφορετικέ καταστάσει. Έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ σωστά στην επιχειρηματολογία των τραπεζών στην Ισπανία όπου πράγματι μετά από μία μείωση ε, του κόστους έκδοσης οι τράπεζες άρχισαν να ζητούν μεγαλύτερα ποσοστά προμήθειας. Να μην ξεχνάμε όμως ε, τι συνέβη τότε όταν οι τράπεζες αύξαναν το κόστος όλων των τραπεζικών προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό ήταν στα πλαίσια μιας κατάστασης όπου ο ανταγωνισμός ε, και οι τράπεζες δεν έπαιξαν ρόλο για να μείνουν τα κόστη χαμηλά. Στη Γαλλία ε, με το λεγόμενο Groupon, Visa και Market και Mastercard ε, δεν επηρεάστηκαν οι αγορές. Στην Ελβετία δεν επηρεάστηκαν οι αγορές. Ε, το κόστος των προμηθειών μειώθηκε στη ΣΥΠΑ μετά από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Οι τράπεζες είχαν ανακοινώσει ότι θα χρέωναν τους καταναλωτές 55 δολάρια το χρόνο τους καταναλωτές και αυτός ήταν άλλωστε και ένας από τους λόγους για τους οποίους τότε ξεκίνησε και το κίνημα αντίδρασης, το λαϊκό κίνημα αντίδρασης Occupy. Ε, είχαν πει ότι αρνούνται τέτοιου είδους ε, ε, κάρτες και στο τέλος απέσυραν τις προτάσεις τους αυτές όλες οι τράπεζες. Όλα εξαρτώνται λοιπόν από τις αγορές, από τις συμπεριφορές των πιστοτικών ιδρυμάτων και από τον ανταγωνισμό. Λοιπόν και τέλος, καινοτομία. Πολύ, πολλές φορές ακούμε τα προγράμματα και τις τράπεζες να λέγουν ότι αν τυχόν δεν μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με αυτά τα κρυφά κόστη δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όλες τις καινοτομίες που είναι απαραίτητες για τις ιντερνετικές πληρωμές, για τις πληρωμές με κινητά κτλ. Ποτέ δεν μπορέσαμε να συνδέσουμε την καινοτομία και αυτά τα κόστη των προμηθειών. Τα κόστη των προμηθειών ήταν υψηλότερα για τις παλαιού τύπου κάρτες ε, όπου έπρεπε να υπογράφει στο ταμείο κάποτε. Δεν ήταν ασφαλή τα συστήματα αυτά, ήταν πάρα πολύ αργά και αναποτελεσματικά και τα συνέχιζαν οι τράπεζες γιατί είχαν υψηλή προμήθεια. Και εκεί λειτουργήσε λοιπόν η προμήθεια εις βάρος των ε, συναλλαγών και της καινοτομίας. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν ε, ε, επενδύσεις αλλά από πλευράς των τραπεζών και των εμπόρων. Ήδη πληρώνουν οι έμποροι και θα πληρώνουν ακόμα περισσότερο αν δεν μειωθούν. Δεν είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι συνδέεται η καινοτομία και οι προμήθειες. Τέλος, πιστεύουμε ότι αν πράγματι θέλουμε να υπάρξει καινοτομία στην Ευρώπη, ας επιλέξει ο καταναλωτής. Να πει ο καταναλωτής αν θέλει να χρηματοδοτήσει ένα τηλέφωνο ή ένα, μια ηλεκτρονική πληρωμή και να μην υπάρχουν κρυφές επιβαρύνσεις και κρυφή φόροι εις βάρος του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας έλειψε καθόλου ειλικρινά η, ε, η διαφάνειά σας. Ήσασταν τόσο σαφείς. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες, ε, απαντήσατε από τις περισσότερες από τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να δευτερολογήσει. Κύριος Μπίλαν, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους ε, για όλα όσα είπαν. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους ιδιαίτερο την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια καταπληκτική παρουσίαση και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα καλύφθηκαν από την παρουσίασή της. Ε, αναμένω λοιπόν καλή συνεργασία με τους ε, σκιώδεις ηγητές ε, για την περαιτέρω πορεία της έκθεσής μου. Το χρονοδιάγραμμα λέει ο Πρόεδρος. Επειδή θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό και από απόψε τους καταναλωτών είναι γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Προθεσμία λοιπόν για τις τροπολογίες 10 Δεκεμβρίου Ελπίζω οι σκιώδεις συζητητές να συναντηθούν πιο πριν ε, για να χωνέψουν μερικές από τις πληροφορίες αυτές. Θα μας στείλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Διαφάνειας για τις οποίες μίλησε, οπότε θα έχετε όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε, ότι, να καταλάβετε ένα πολύ δύσκολο και περίπλοκο θέμα. 22 και 23 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες ε, και στις 10 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ, από ό,τι κατάλαβα, θα ε, ψηφίσουν στις 20 Φεβρουαρίου και θα δούμε και τι θα κάνει και η Ελληνική Προεδρία με το θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα σημειωθεί γρήγορη πρόοδο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ την κυρία Βέιζενμπεκ και την ομάδα τη, όλο ιδιαίτερο. Ε, ελπίζω να είστε εδώ όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Τρεις η ώρα θα ξανααρχίσει η συνεδρίασή μας το απόγευμα και θα υπάρξει και ακρόαση για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. εισηγητή ο υποφαινόμενο. Θα έχουμε πάρα πολύ καλού ομιλητέ, πολύ καλή για ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τρει η ώρα ακριβώ λοιπόν το απόγευμα και ο κύριο Κοφεράτη θα είναι ο πρόεδρο ώστε εγώ να ασκήσω την ιδιότητα του εισηγητή και να κάνω ερωτήσει. Θα σα δω λοιπόν στι τρει η ώρα ελπίζω και ευχαριστώ και πάλι όλου σα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.